Um, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε σήμερα το πρωί με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές για σήμερα το πρωί. Το σημείο 16, όπως βλέπετε, έχουμε ε, μαζί μας τον Επίτροπο Δημήτριο Αβραμόπουλο, που είναι ο Επίτροπος Αρμόδιος για την Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ιθαγένεια. Ε, θα μας μιλήσει για την εμβεβαιότητα θεωρήσεων Οπότε 9 ναι, με 11 θα λάβει χώρα η ακρόαση αυτή και όχι στις 11 όπως είχαμε προβλέψει. Στα σημεία 3 με 10 θα λάβουν χώρα 11 με 12. Θα το δείτε και στο νέο πρόγραμμα. Το σημείο 22 θα εξεταστεί στις 10 πριν από το σημείο 21 και το σημείο 23 που είναι η παρουσίαση του σχεδίου αποστολής ε, ε, τη έκθεση αποστολή που έγινε στο Καλέ αναβάλλεται για την επόμενη φορά. δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται. Όσον αφορά το γλωσσικό, δυστυχώς τα κρατικά, τα μαλτέζικα και τα γκέλικ δεν είναι διαθέσιμα σήμερα. Τώρα, συστάσεις των συντονιστών βάσει του άρθρου 205. Πρώτα απ' όλα ορίζονται εισηγητέ. Ο κύριος Χάλα Άχο, το ICR, ορίστηκε εισηγητής για τον προτινόμενο κανονισμό όσον αφορά την ενιαία μορφή που θα έχουν οι άδειε διαμονής. Ε, Συντάκτε γνωμοδοτήσεων. Ο κύριος Γέζεκ από την άλλη ορίστηκε συντάκτης γνωμοδότησης για τις απαλλαγές για το έτο 2015 όσον αφορά τη Europol, τη Eurojust, τη Frontex, την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την MCDA, ΣΕΠΟΛ, ΆΣΟ κλπ. Ε, εγκρίνεται τις ε, συστάσεις αυτές των συντονιστών. Μάλιστα. Επίσης, θα έχουμε μια σύντομη ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 10.40. Οπότε παρακαλώ να έχετε τις ηλεκτρονικές σα κάρτες ψηφοφορίας. Ωραία, αν είμαστε έτοιμοι, α περάσουμε στην ημερήσια διάταξη αυτή καθ' αυτή, που αρχίζει με το σημείο 16, όπως σας είπα. Και πολύ χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον ε, Επίτροπο Δημήτριο Γραμμόπουλο. Θα έρθει και σήμερα το απόγευμα στην ακρόαση που θα έχουμε για το Σέγγελ. Και είναι καλό που θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να μιλήσουμε περισσότερο επί της ουσίας για αυτά. Πάντως προς το παρόν, Δημήτρη, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας το σημαντικό αυτό θέμα της αμοιβαιότητας θεωρήσεων. Όπως γνωρίζετε, οι πολίτες διαφόρων χωρών μελών χρειάζονται θεωρήσει για να μπαίνουν στον Καναδά ή τις Ηνωμένες ενώ οι πολίτε των χωρών αυτών δεν χρειάζονται θεωρήσει για να μπαίνουν στον χώρο Σέγγεν. Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό και πήγει για μα. Οπότε θα σας υπενθυμίσω τι συζητήσει είχαμε κατά το παρελθόν από αυτά. Στι 12 Απριλίου φέτος εγκρίναμε μια καταξιδότηση πράξη που προβλέπεται στον κανονισμό 53901 σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση που συζητήθηκε στην Επιτροπή μας στις 20 Απριλίου. Στη συνέχεια και βάσει της απόφασης των συντονιστών της ΛΥΜΠΕ της 10ης Μαΐου, στις 7 Ιουνίου έγραψα στον Επίτροπο Αβραμόπουλο και του είπα ότι θεωρούμε υποχρέωση κατά τη γνώμη μας, να υιοθετηθεί η καταξιδότηση πράξη στον κανονισμό 539 κάθετος 2001 όσον αφορά την άρση της κατάργησης θεωρήσεων για υπηκός τρίτων χωρών. Ορισμένο τρίτο χωρών. Στις 13 Ιουλίου η Επιτροπή παρουσίαζε μια επιπλέον ανακοίνωση όσον αφορά την σημερινή κατάσταση για την μία αμοιβαιότητα στα θέματα θεωρήσεων και παρουσιάστηκε στη Λίπε στις 31 Αυγούστου από τον κύριο Ολιβιέ Ονίδη, που είναι πληρωτής Γενικός Διευθυντής της DG Home. Στις 13 Σεπτεμβρίου οι συντονιστές Λίμπε την παρουσία του προηγούμενου εισηγητή μας για αυτά τα θέματα, του κυρίου Ντίεθ Ντεμέρα, αποφάσισε να καλέσουμε τον Επίτροπο Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να συμφωνήσει και να έρθει εδώ σήμερα. Οπότε θα ζητήσω από τον Επίτροπο να σχολιάσει τα θέματα αυτά και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντίαθ Ντεμέρα και σε οποιαδήποτε άλλον επιθυμεί να πάρει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ και σας παρακαλώ σχολιάστε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. you, uh, Ευχαριστώ, Κλοντ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Θα αρχίσω ευχαριστώντας σας για άλλη μια φορά που με φέρατε εδώ προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτά τα σημαντικά θέματα που είναι πονοκέφαλος για μένα, μεγάλος. Αλλά τι να κάνουμε. Με τη βοήθειά σας θα βρούμε διέξοδο. Για το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και εκτιμά ιδιαίτερα που έχουμε διάλογο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι συμφωνούμε όλοι πως πρόκειται για ένα πολύ το ζήτημα. Το θέμα της αμοιβαιότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Έχει να κάνει αφενός, η αμοιβαιότητα δηλαδή, με την έλευση διακρίσεων σε βάρος των Ευρωπαίων πολιτών, αφετέρου όμως έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό που εννοώ είναι ότι δίνουμε προτεραιότητα στη στρατηγική μας να πετύχουμε την ε, λύση του ζητήματος αντί να πούμε σε μία σύγκρουση που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για όλες τις πλευρές. Αντιλαμβάνομαι πλήρω τι δικέ σα προσδοκίε, να υπάρξουν δηλαδή απτά αποτελέσματα και πρόοδο. Γι' αυτό λοιπόν θα αρχίσω με τον Καναδά. Γνωρίζετε τις προσπάθειες που έχω κάνει, γιατί και για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό. Υπήρξε μια σαφής ευκαιρία για επικοδομητικό διάλογο. Γνωρίζετε ότι το θέμα αυτό συνδέεται με την Βουλγαρία και την Ρουμανία όσον αφορά την εμπορική συμφωνία και την συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Η υπογραφή των συμφωνιών αυτών είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα έχουμε στη διάσκεψη κορυφής με τον Καναδά που θα λάβει χώρα στις 27 Οκτωβρίου. Η συζήτηση έγινε σε αυτό το πολιτικό επίπεδο πριν από λίγο καιρό. Συναντήθηκα με τον κύριο Μακάλουμ που είναι ο Καναδός ο Υπουργός για να διαπραγματευτούμε επί μιας λύσης. Τον Ιούλιο, για πρώτη φορά, ο Καναδάς υποσχέθηκε να προσφέρει χρονοδιάγραμμα για την άρση της υποχρέωσης ε, θεωρήσεων. Τώρα λοιπόν είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε αυτό. Έντονος διάλογος λαμβάνει η χώρα με όλους τους εμπλεκόμενους, με όλες τις πλευρές, στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν λύσεις που προτείνονται πάνω στο τραπέζι και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Η πρόοδος που βλέπουμε με τον Καναδά δείχνει ότι η προσέγγιση μας ήταν η ορθή. Διπλωματία δέσμευση από όλες τις πλευρές είναι πράγματα που φέρουν αποτελέσματα. Η άρση αυτής της υποχρέωσης πιστεύω ότι θα προχωρήσει και είμαι ουσιαστικά σίγουρος ότι εάν βάζαμε εμείς θεωρήσεις για τους Καναδούς, αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Έρχομαι τώρα στις Ηνωμένε Πολιτείες συνεχίζουμε τις συζητήσεις με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Δεν μπορώ να πω ότι σε αυτό το στάδιο έχουμε πρόοδο. Όπως κάνω πάντα, θα είμαι και πάλι εδώ σήμερα ειλικρινής μαζί σας. Πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές στο Κογκρέσο, δεν αναμένω αλλαγή. Και αντιλαμβάνεστε γιατί. Είναι επίσης περιττό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι το θέμα αυτό το κρατάμε πάνω-πάνω στους στόχους μας για να το συζητήσουμε με τη νέα κυβέρνηση και το Κογκρέσο. Δεν είναι θέμα έλλειψης βούλησης να φέρουμε σε πέρα στις υποχρεώσεις μας ή να υποστηρίξουμε κάτι το οποίο είναι δίκαιο. Το θέμα είναι το πότε θα το κάνουμε αυτό, να επιλέξουμε την πιο κατάλληλη στιγμή για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε. Η στρατηγική μας είναι η ίδια όπως και με τον Καναδά. Αντί δηλαδή να παίρνουμε αντίπεινα που είναι αντιπαραγωγικά, επιλέγουμε την δέσμευση, την παρακολούθηση και όπως σας είπα υπομονετική διπλωματία. Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών παίζει ζωτική σημασία ρόλο σε αυτή την υπόθεση δεν μπορεί να υπάρξει επέκταση του προγράμματος χωρίς να υπάρξουν νομοθετικές αλλαγές. Το σημερινό Κογκρέσο απλώς δεν θα δεχότανε να αλλάξει το πρόγραμμα αυτό άρσης της υποχρέωσης θεώρησης για τις εναπομείνουσες πέντε χώρες μέλη. Συνεχίζουμε να θέτουμε το ζήτημα πάντως και εσείς να το κάνετε κάθε φορά που συναντιέστε με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου γιατί πρόκειται για μια κοινή μεταξύ μας προσπάθεια. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η Επιτροπή δεν θα διστάσει να εγκρίνει τις πράξεις που χρειάζεται αν γνωρίζαμε ότι αυτό θα οδηγούσε στην άρση θεωρήσεων για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Όμως για τις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουμε σίγουρα ότι η επίπτωση θα ήταν ακριβώς το αντίθετο από το επιθυμητό. Δηλαδή ακόμα και η έγκριση μιας κατεξοδότηση πράξης από την Κομισιόν θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρο αυτό το πρόγραμμα άρση της υποχρέωσης θεωρήσεων ε, με τις ΗΠΑ και θα οδηγούσε κατά πάσα πιθανότητα στην εκ νέου εισαγωγή της υποχρέωσης θεώρησης για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που θα ταξίδευαν προς τις ΗΠΑ. Οπότε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που έχει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις αρνητικές συνέπειες που θα είχαν οι κανόνες μας. Συνέπειες οι οποίες θα γινόντουσαν αισθητέ στους πολίτες μας και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη στρατηγική σημασία σχέσεις μας. Εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε συχνά μαζί σας και να συζητούμε τα αποτελέσματα των προσπάθειών μας. Θέλουμε βεβαίως αμοιβαιότητα για το θέμα της θεώρησης για όλες τις χώρες μέλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το θέμα σήμερα μαζί σας. Ευχαριστώ Δημήτρη. Αρκετοί συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο το οποίο είναι κατανοητό, είναι πολύ σημαντικό και λεπτό θέμα. Θα αρχίσουμε με τον πρώην εισηγητή, κύριο Ντίαθ Ντεμέρα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και εσάς, κυρία Βραμόπουλε, που ήρθατε εδώ ε, ενώπιον της Επιτροπής μας. Και επειδή κρατάτε ε, σταθερή στάση και επιμένετε ενώπιον ενό τόσο περίπλοκου ζητήματο. αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα και εκτιμώ και την ειλικρίνεια των λόγων σας. Ε, επειδή λοιπόν είστε τόσο ειλικρινείς, θα ήθελα να ακούσετε κι εσείς με ειλικρίνεια τη θέση του εισηγητή, που είναι βασικά και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως γνωρίζετε κύριε Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση είναι επανάληψη των όσων είπαμε στις 20 Απριλίου και 31 Αυγούστου. Ε, τότε η Κομισιόν δεν έχει αλλάξει την θέση της. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, ωστόσο είναι εξίσου αλήθεια ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαφώς μία... Ε, δυσκολία ε, μια ατελή διαδικασία. Καταλαβαίνω, κύριε Βραμόπουλε, πολύ καλή πέρα από τις εξηγήσεις που μας δώσατε σήμερα, που είναι ελπιδοφόρες στην περίπτωση του Καναδά, αλλά απογοητευτικές στην, για την ΕΠΑ. Ελπίζω λοιπόν ότι θα ασκήσετε μια πολύ ισχυρή διπλωματική πίεση, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην νομιμότητα. Είναι μια συζήτηση που αφορά όχι την ουσία αλλά την τήρηση της νομοθεσίας. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε αν θα είναι σωστό ή όχι να φέρουμε την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες των ΗΠΑ ή του Καναδά. Ωστόσο, θα πρέπει να ε, τηρηθεί νομοθεσία 539 2001. Ε, σύμφωνα δηλαδή με την απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο ενεργεί με υπευθυνότητα και από τον ε, Μάιο κάναμε δύο συζητήσεις στην Επιτροπή, δύο συζητήσεις στους συντονιστές και μία διμερή συζήτηση που είχα την ευκαιρία να έχω εγώ με τον ε, Επίτροπο. Εγώ σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας κύριε Αφραμόπουλε, για τις ενέργειες τις οποίες προβαίνει η Κομισιόν ώστε να ε, τηρηθεί η αμοιβαιότητα με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το αποτέλεσμα των διμερών συζητήσεων που και εσείς είχατε τα τελευταία, τις τελευταίες εβδομάδες είναι πολύ σημαντικά. Ε, επαναλαμβάνω και δεν θα πάψω να επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να συνεχίσετε να πιέζετε στο πλαίσιο των διπλωματικών σχέσεων ε, με τις χώρες αυτές ώστε να εξευρεθεί λύση σε αυτή την υπόθεση. Όμως ταυτόχρονα παραλλήλως θα πρέπει να τηρηθεί και το αρθρο 1.4.F του κανονισμού που υποχρεώνει την Κομισιόν να παρουσιάσει κατεξιδότηση πράξη εφόσον έχουν περάσει 24 μήνες από την ε, ε, κοινοποίηση της έλλειψης ε, αμοιβαιότητας. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να γίνει και αυτό το έχει επιβεβαιώσει και το ΔΕΚ στην απόφασή του της 16ης Εβδόμου του 2015. Δεν ναι, λέει πουθενά ότι η Κομισιόν θα πρέπει, αν θα πρέπει να παρουσιάσει δύο, μία ή δύο ανακοινώσεις. Όχι. Ε, Δεν σας κρύβω ότι είναι λογική αυτή η διαδικασία, αλλά περίπλοκη και η Κομισιόν όμως έτσι διοποιείται αρμοδιότητες που δεν έχει, που δεν είναι δικές της κανονικά. Ε, επεμβαίνει δηλαδή στις ε, αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και αδιαμφισβήτητα ε, βρισκόμαστε ενώπιον ενό διαθεσμικού προβλήματο και είναι απαραίτητο η Κομισιόν να ενεργήσει Ω πραγματικό θεματοφύλακα των συνθηκών. πέραν αυτής τη κατάστασης ζητώ από τον κύριο Επίτροπο με κάθε καλή θέληση και ταπεινότητα ε, και σεβασμό. Σας ζητώ λοιπόν κύριε Επίτροπε να σεβαστείτε τον κανονισμό, να παρουσιάσετε, να υποβάλλετε την καταξιδότηση πράξη και τότε εμείς μαζί με το Συμβούλιο, οι συνομοθέτες, θα συζητήσουμε όσον αφορά την καταλληλότητα και τις πολιτικές συνέπειες μιας πιθανής επανεισαγωγής των θεώρησης και θα αποφασίσουμε τι να κάνουμε. Όμως αυτή είναι απόφαση που αναλογεί σε εμά ως συνομοθέτες. Αναλογεί σε εμά και στο Συμβούλιο. Διαφορετικά, τι δρόμος μας μένει για να τηρηθεί η νομοθεσία. Ένας είναι ο δρόμος, αλλά ε, δεν θέλω καν να το αναφέρω. Να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι εγώ είμαι φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν επιθυμώ την επιβολή θεωρήσεων στους πολίτες αυτής της σπουδαίας χώρας, όμως αυτό που επιθυμώ πάνω απ' όλα είναι ότι τόσο ο Καναδάς όσο και η ΕΠΑ ε, να εφαρμόσουν την άρση των θεωρήσεων για την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Κύριε Αβραμόπουλε, μην πιστεύετε ότι, μην πιστέψετε ότι δεν εκτιμώ τη δουλειά σας. Αντιθέτως, την εκτιμώ πάρα πολύ. Και εκτιμώ ότι πρέπει να υπάρχει αρμονία ανάμεσα στη στρατηγική και την αποτελεσματικότητα. Όμως ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λάβετε υπόψη πόσο αποτρεπτικό θα ήταν για απέναντι στην αντίσταση του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών να αποφασίζαμε εμείς ενώ μετά από την ε, πράξη ε, την κατεξοδότηση να επιβάλλουμε θεώρηση στο υπόλοιπο το, και των κρατών μελών. Και γι' αυτό θα είχαμε αντίθετο. Το, θα έπρεπε να κινηθεί τόσο και το Κογκρέσο. Εξαίρεση για τις θεωρήσεις των πέντε χωρών, αλλά και για την επαν, επανεισδοχή των θεωρήσεων για τις, όλες τις χώρες της Ένωσης. Δεν ήταν αυτό ένα βολικό στρατηγικό μέσο ώστε να μπορέσουμε να, να, να αναγκάσουμε το Κογκρέσο τον ΗΠΑ να κινηθεί από νομικής πλευράς. Τώρα, συνέπειες βέβαια, θα πρέπει να τις ε, εκτιμήσουμε σωστά. Όμως η Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν είναι ένα βασικό ε, πυλώνας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ε, αυτή πρέπει να αποφύγει τις ζημιές και τις συνέπειες. Και η Κομισιόν είναι αυτή που πρέπει να εγγυηθεί την εφαρμογή του νόμου για την οθεματοφύλακα των συνθήκων. Ήδη το είπα και το είπαμε και το λέμε και στη γλώσσα μου ότι είναι η καυτή πατάτα. Το ποιος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα που λέμε εμείς ε, στα ελληνικά. Η Κομισιόν πρέπει να τηρήσει τον κανονισμό αυτόν ε, που ισχύει και βέβαια θα πρέπει να κάνει ένα πάρα πολύ δύσκολο διπλωματικό έργο. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Είναι, ήσασταν σαφής από την πλευρά του Κοινοβουλίου, μάλιστα. Η κυρία Ζίπελ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων στον κύριο Ντία Στεμέρα για την πλήρη ανάπτυξη του θέματος και συμφωνώ απολύτως με τα όσα δήλωσε σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις. Γι' αυτό θα μπορέσω να είμαι σύντομη, διότι Ήδη είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη σχετικά με το ποια μηνύματα δίνουμε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα. Έχουμε μια ξεκάθαρη συμφωνία μεταξύ άλλων με τον Καναδά και με τις Ενωμένε Πολιτείε με ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την διευκόλυνση, για, την, για να καταστεί δυνατή δηλαδή ε, μετακίνηση χωρίς προξενικές θεωρήσεις. Και κανείς δεν ήταν τηρεί αυτά τα πράγματα. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διστάζει μεταξύ άλλων να εκδώσει την κατεξουσιοδότηση πράξη, διότι βεβαίως μπορεί αυτό να έχει επιπτώσεις. Και όπως είπε ο Δίας Τεμέρα, δεν θέλουμε στην πραγματικότητα να απαιτήσουμε προξενικέ θεωρήσει για όλου του Αμερικανού πολίτε, αλλά και για του Καναδού ενδεχομένω. Δεν ξέρουμε αν τούτο το μήνα θα υπάρξει συμφωνία άλλωστε. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί φαίνεται πω είναι λιγότερο διστακτικοί. Δηλαδή, οι ίδιοι δεν τηρούν τι δεσμεύσει του και έρχονται και μας απειλούν από πάνω ότι θα επιβάλλουν προξενικές θεωρήσεις, υποχρέωση δηλαδή έκδοση προξενικών θεωρήσεων, για τους πολίτες και των 28 χωρών μελών. Α, και εμείς λέμε, όχι, ίσως είναι επικίνδυνο να αντιδράσουμε. Εάν βλέπω εγώ τέτοια πράγματα, εγώ τουλάχιστον ω Αμερικανικό Κογκρέσο ή Αμερικανική κυβέρνηση θα έλεγα, μα ποιο μπορεί να του πάρει σοβαρά του Ευρωπαίου. Ακόμη και αν εμείς, δηλαδή οι Αμερικανοί, δεν τηρούμε τι υποχρεώσει μα, δεν έχει απολύτω καμία συνέπεια. Θεωρώ λοιπόν ότι ο τρόπος που αντιδρούμε έχει συνέπειες όχι μόνο στην αμοιβαιότητα του, του καθεστώτος προξενικών θεωρήσεων, είναι και ζήτημα εμπιστοσύνης στην συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνει το βήμα, να εκδοθεί δηλαδή η κατεξουσιοδότηση πράξη και να πράξουμε πάντα το δυνατό ώστε εν τέλει να υπάρχει αμοιβαίως ελευθερία θεωρήσεων και από τις δύο πλευρές, Αμερικανούς, Καναδούς και τις 28 χώρες μέλη της Ένωσης. Να μην χρειαστεί να περάσουν άλλοι 6 μήνες, ούτε ακόμα χειρότερα 2 ή 3 χρόνια. Αλλά πρέπει αυτά να γίνουν σχετικά σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία... Ευχαριστώ ευχαριστω ευχαριστω πολυ τα τελευταία δύο χρόνια Σχετικά με τον κανονισμό 1289 του 13, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί την κατάσταση σχετικά με την έλλειψη αμοιβαιότητος σε ό,τι αφορά τα καθεστώτα προξενικών θεωρήσεων. Πρόκειται για μια κατάσταση που επηρεάζει εκατομμύρια πολιτών σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Πολωνία και άλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται ότι οφείλει να αναλάβει δράση. Δηλαδή θα πρέπει να εκδώσει την κατεξουσιοδότηση πράξη. Ανταυτού στι 12 Τετάρτου φέτος, όταν δηλαδή έληξε η προθεσμία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μετακυλήσει το καθήκον αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ο κανονισμός, ωστόσο, λέει καθαρά στις διατάξεις του και ο πρόεδρος μας Κλοντ Μωράης το είπε ήδη, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εκδώσει την κατεξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την έλλειψη απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων, έχοντας υπόψη ότι η αντίστοιχη τρίτη χώρα δεν έχει άρει την υποχρέωση προξενικών θεωρήσεων εντός του 24 μήνου. Και επαναλαμβάνω, η προθεσμία έληξε στις 10 Απριλίου του 2016. Η ερώτησή μου είναι πώς νομίζετε ότι θα αντιδράσουν, θα το, πώς θα το εκλάβουν οι, οι, οι Ευρωπαίοι πολίτες, ιδίως των χωρών που θίγονται. Και τι κάνει αυτό. Τη ζημιά κάνει αυτό στο κύρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε την αίσθηση πλέον ότι ζούμε σε μια Ευρώπη δύο διαφορετικών κατηγοριών πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν απειλεί ότι θα πράξει κάτι το οποίο δεν πράττει ποτέ. Υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Κάνει όμως άλλα πράγματα, αντί να προβάλλει, να προωθήσει αυτά που επιθυμεί και θέλει και πρέπει να προσπίζεται. Είστε και όσοι έπρεπε να το είχα πει από πριν. Η κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο για την δέσμευσή του στο θέμα και για την συνεκτική πολιτική την οποία ακολουθεί και εφαρμόζει σε συνεργασία με τις χώρες μέλη τους τελευταίους μήνες στην προσπάθεια να επιτύχει την αμοιβαιότητα στο καθεστώς προξενικών θεωρήσεων. Η άρση της υποχρώσεως για έκδοση προξενικών θεωρήσεων είναι σημαντική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω βεβαίω για τη χώρα μου, τη Βουλγαρία. Διότι οι Βούλγαροι πολίτε εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να ζητούν έκδοση προξενική θεωρήσεω για να πάνε στην ε, Αμερική, δηλαδή στι ΗΠΑ ή στον Καναδά. Έχουν γίνει ε, ξεκάθαρες δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Μάρκον ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Εγώ επιθυμώ να πω το εξή. Φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα ήδη. Τον περασμένο μήνα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργό συνομίλησε με τον Καναδό Πρωθυπουργό κύριο Τριντό. Ο Καναδάς ήδη προχωρεί την διαδικασία για την άρση της υποχρέωσης θεωρήσεων για τους ε, Βουλγάρους πολίτες και τον Φεβρουάριο του επομένου έτους θα δέχεται ο Καναδάς Βούλγαρους πολίτες να επισκέπτονται την επικράτειά του χωρίς ε, προξενικές θεωρήσεις. Και κάποιο διάστημα, αυτό σε μια πρώτη φάση για όσους έχουν ήδη ταξιδέψει ή για όσους έχουν αμερικανικές ε, προξενικές θεωρήσεις. Και αργότερα θα ισχύσει αυτό για όλους τους Βουλγάρους πολίτες. Υπάρχουν βεβαίω ορισμένε τεχνικέ δυσχέρειε, καθώ και διοικητικού χαρακτήρα, που ίσω οδηγήσουν σε κάποια αναβολή μέχρι τις 18 Πέμπτου 2000, όχι με συγχωρειτε Μαΐου μάλλον, 1η Πέμπτου 2018. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ήδη να διαγράφονται κάποια ξεκάθαρα αποτελέσματα. Και αυτά όντω οφείλονται στι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή οι Βούλγαροι πολίτε πραγματικά βλέπουν κάποια αποτελέσματα. Ε, επισημαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην προκαλέσουμε στο κοινό την εντύπωση ότι η Ευρώπη κινείται με δύο διαφορετικέ ε, ε, ταχύτητες και ότι δημιουργούνται δύο διαφορετικέ κατηγορίε πολιτών. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι σύντομα και απτά. Η ερώτησή μου έχει ως εξή. Πιστεύετε ότι τα όσα έχουμε επιτύχει ως τώρα με τον Καναδά μπορούν να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε περαιτέρω στο ίδιο θέμα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει η συμφωνία με τον Καναδά ως μοντέλο και για αυτό, αυτήν με τους Αμερικανούς. Ευχαριστούμε. Κυρία Κάμπριελ, ο κύριος Σαλχάου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ποιε είναι οι απαιτήσει των Ηνωμένων Πολιτειών για τι πέντε χώρε. και οι απαιτήσει αυτέ θα προχωρήσουν για τις πέντε αυτές χώρες, θα μπορέσουν δηλαδή να τις καλύψουν αυτές οι πέντε χώρες σύντομα. Μπορώ να συμφωνήσω με τον Επίτροπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μια αντιπαράθεση με τις Ηνωμένε Πολιτείες δεν είναι καθόλου σοφή, καθόλου καλή ιδέα και είναι μάλλον αντιπαραγωγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως είναι ένα ετερογενές σώμα χωρών. Οπότε ακόμα και αν παριστάνουμε ότι δεν ισχύει αυτό, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μας βλέπουν ως ένα ετερογενές σώμα. Πάντως, τι εικόνα δημιουργείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις άλλες χώρες. Θα έπρεπε βέβαια να αναρωτηθούμε τι ζημιά ε, θα υπήρχε στην, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις υπόλοιπες 23 χώρες αν και αυτές χάνανε το σύστημα εξαίρεσης από την υποχρέωση θεώρησης. Πρέπει και αυτό να το σκεφτούμε. σε ευχαριστώ. Άλλοι δύο, Βίλστρομ και Ράντεβ και κλείνω τον κατάλογο μιλητών. Η κυρία Βίλστρομ έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ, Σεσίλια. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα το πρωί. Αισθάνομαι ότι επαναλάβατε αυτά τα οποία μας είπατε και πριν από ένα μήνα. Και δεν υπάρχει πρόοδος. Αυτή η διπλωματική προσέγγιση ποια είναι, όταν ξέρουμε ότι αυτό που θα πρέπει να έχουμε είναι πλήρη συμμόρφωση προς τον κανονισμό, ιδιαίτερα το άρθρο 1.4f, αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να προχωρήσει σε κατεξουσιδότηση πράξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνω το λόγο που λέτε ότι διπλωματικά προσπαθείτε να πετύχετε αποτελέσματα, αλλά δεν υπάρχουν αποτελέσματα μέχρι τώρα. Και συμφωνώ και με αυτά που είπε ο εισηγητής και είμαι περήφανη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να έχει ευρωβουλευτές όπως ο συνάδελφος Δίεθ που ακολουθούν τις αρχές τους, που υποστηρίζουν το σώμα αυτό, που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενότητά της και τους πολίτες στις πέντε χώρες. Γιατί ε, αυτές οι χώρες θα τον δούνε σαν ήρωα τον κύριο Δίεθ Δεμέρα, ο οποίος υποστηρίζει ξανά και ξανά τα δικαιώματά τους Πράγμα το οποίο φαίνεται να μην κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί δεν το κάνει. Γιατί εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα κάνουμε λιγότερα από όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε μια μεγάλη οικονομία, ισχυρή. Γιατί πρέπει πάντα εμείς να παρετούμεθα από τα δικαιώματά μας ξανά και ξανά και ξανά. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τώρα, από νομική άποψη. Εμείς από νομική άποψη βρισκόμαστε απέναντι σε μια κατάφορη αποτυχία δράσης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ανέλαβε δράση και θα έπρεπε να έχει νομικές συνέπειες αυτό. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δράσει κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τηρώντας πλήρως όλες τις συνθήκες. Ελπίζω και επιθυμώ να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Επιθυμώ να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι διακυδεύονται τόσα πολλά πράγματα, συμφωνίες με τις Ηνωμένε Πολιτείες, μιλάμε για τη συμφωνία TTIP, Είμαστε δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο. Αν δεν υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, τότε τι θα γίνει στο μέλλον και σε μελλοντικέ συμφωνίες για το εμπόριο. Πιστεύω λοιπόν από βάθος καρδίας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να σταματήσει να εκδίδει ανακοινώσει και να αρχίσει τη δράση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Να αναλάβει δηλαδή τη νομική ευθύνη και να φέρει αποτελέσματα. Και το ξαναλέω. Πρέπει να νιώθουμε ελεύθεροι να δράσουμε. Δεν είμαστε εμείς υποτακτικοί κανενός, όχι επειδή μας πιέζουν να μην κάνουμε τίποτα. Είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να υπάρξει συμφωνία. Η αμοιβαιότητα πρέπει να ισχύσει. Φανταστείτε εμείς να αποκλίναμε πέντε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτές σαν να πρόκειται για πολιτείες δεύτερης κατηγορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνώ απόλυτα με τη φίλη από αυτού. Πρέπει να δείξουμε στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες και τους πολίτες τους ότι τις ανησυχίες τους τις παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Και για να τελειώσω με μια νότα ελπίδας κύριε Αβραμόπουλε, κινηθείτε. Αυτή είναι η έκκληση που κάνω σήμερα το πρωί, μαζί με τον εισηγητή. Κινηθείτε, αναλάβετε την ευθύνη και φέρτε αποτελέσματα. Δεν θέλουμε πια ανακοινώσεις ούτε επαναλήψεις των ίδιων και των ίδιων. Πρόεδρος, ευχαριστώ Σεσίλια. Ο κύριος Ράντεπο τελευταίος και μετά θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμε Επίτροπε. Πράγματι, οι διπλωματικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντικές. Όμως, έχουν πάρει πάρα πολύ χρόνο. Πράγματι, υπάρχει κάποια πρόοδος όσον αφορά τις σχέσεις μας με τον Καναδά την προηγούμενη εβδομάδα. Για παράδειγμα, ο Βουλγάρος Πρωθυπουργός ε, είχε πληροφορίες από τον Καναδό ομολογό του για το θέμα των θεωρήσεων ότι σιγά σιγά θα υπάρξει η κατάργηση από το 2017 και ότι θα είναι πλήρης η κατάργηση αυτή θεωρήσεων για τους συμπατριώτες μου το 2018. Αλλά αυτή την πληροφορία δεν την επιβεβαίωσε η Επιτροπή. Όσον αφορά το πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων για τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, μετά τις εκλογές, μια νέα κυβέρνηση στις Ηνωμένε Πολιτείες μπορεί να επιτευχθεί κάποια πρόοδος. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα όμως που βλέπετε εσείς προκειμένου να ξέρουμε ποια θα είναι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε αυτό το ζήτημα των θεωρήσεων και της αμοιβαιότητας. Ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σημάδι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τους λέει ότι τελικά οι συμφωνίες μαζί τους είναι πιο σημαντικές από την αμοιβαιότητα και την ίση μεταχείριση όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Μα δεν πιστεύετε εσείς ότι είναι πιο σημαντικό να τηρείται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αντί να βάζουμε προτεραιότητα στις καλές σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η αλληλεγγύη και η αμοιβαιότητα θα έπρεπε να υπερισχύει. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, το περιμένατε βέβαια ερχόμενος εδώ να τα ακούσετε αυτά. Δεν ξέρω όμως αν περιμένατε το συναδέρφους να είναι τόσο ακριβείς και να μιλούν με τέτοιο ενθουσιασμό για το θέμα. Έχουμε συζητήσει και στους συντονιστές με τον κύριο μέρα και με τους άλλους και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Είπατε στην αρχή ότι ελπίζεται η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να συνεχίζει να το θέτει. Λοιπόν, με κάθε σεβασμό το δείξανε και οι ευρωβουλευτέ μα ε, σήμερα πόσο αποφασισμένοι είμαστε ότι όντω το κάνουμε. Όταν πήγαμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, είχαμε πολύ έντονη ανταλλαγή απόψεων με το Υπουργείο Εξωτερικών εκεί. Κατάλαβαν ότι δεν θέλουμε να έχουμε δεύτερης κατηγορίας πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, τα καταλαβαίνω αυτά που λέτε, Καταλαβαίνω το πώς μας βλέπουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά η Επιτροπή μας, η ΛΥΜΠΕ, να ξέρετε ότι έκανε ό,τι περνάει από το χέρι της για να πιέσει για μια υποχρέωση που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε ακούσατε την άποψη όλων των πολιτικών ομάδων εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν υπάρχει πια καμιά αμφιβολία για το ποια είναι η στάση μας. Για μας είναι υποχρέωση να προχωρήσουμε στην πολιτική πίεση. Οι συνάδελφοι θέλουν να δουν αν συμφωνείτε. Ήθελα να το πω πριν απαντήσετε εσείς. Για να ξέρετε και να ξέρετε επίσης ότι θα προχωρήσουμε και σε προφορική ερώτηση. Είναι σημαντικό για μας η διαδικασία Οπότε, σας παρακαλώ να απαντήσετε. <coughs> Ευχαριστώ, Κλοντ. Ναι. Δεν είναι με ένα έκπληξη, αλλά δεν περίμενα κιόλα ότι θα είμαι το ευπρόσδεκτος εδώ. Είμαι πάρα πολύ ρεαλιστής και έμπειρος πολιτικός. Εγώ σας ζητώ να προσεγγίσετε το θέμα από πολιτικής άποψης, όχι από θεωρητικής ή νομικής άποψης. Και αυτό προσπάθησα να κάνω και εξ αρχής με τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Ε, αγαπητοί φίλοι ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τα όσα είπατε και θα πρέπει να σας πω ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας για την κατάσταση. Ε, και εγώ ανησυχώ, είναι, έχω με τις ίδιες τον ίδιο προβληματισμό. Όλοι θέλουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα πλήρες, πλήρη, πλήρη αμοιβαιότητα θεωρήσεων για τους πολίτες μας που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Όλους μας τους πολίτες. Επίσης γνωρίζουμε ποιες, ποιες, είναι οι, ποιες είναι οι νομικές μας υποχρεώσεις και όπως είπαμε η Κομισιόν είναι νομοταγές ε, θεσμικό όργανο. Όμως Πιστεύω ότι αν ε, παγώναμε τι διαπραγματεύσει δεν θα πετυχαίναμε τίποτα. Δεν είναι προ το συμφέρον οποιοδήποτε από του θεσμού να πάει στο δικαστήριο κατά του άλλου. Δηλαδή να αρχίσουμε να ζεκωνόμαστε στο δικαστήριο για αυτό το θέμα μεταξύ μα. Αυτό δεν θα οδηγήσει σε πλήρη άρση το να θεωρήσουν ούτε για τη ΣΥΠΑ ούτε για τον Καναδά. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα διαπραγματικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πολιτικός μας ε, στόχος με τον Καναδά ε, μάλλον θα φέρει αποτελέσματα σύντομα. Αυτό που σας ζητώ είναι λίγη περισσότερη υπομονή. Με τη ΣΥΠΑ πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας τώρα και μετά από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Είμαστε όλοι πολιτικοί. Ξέρετε ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί εκεί. Πώς... Ξέρετε τι γίνεται με τις εκλογές. Ε, ε, σας καλώ λοιπόν να μας στηρίξετε σε αυτή την προσπάθεια. Η τρέχουσα κατάσταση στις θα επανέλθω σε αυτό με τις εκλογές εκεί τώρα. Δεν μας δίνουν πολλές πιθανότητες για επιτυχία. Θα είμαι σαφής, θα είμαι ξεκάθαρος. Η μόνο η έγκριση εν μιας κατεξοδότηση πράξης ε, θα οδηγούσε αμέσως, ακόμα και πριν να προλάβει να υιοθετήσει θέση το Ευρωκοινοβούλιο, σε ακύρωση αναστολή μάλλον της, ε, ε, της ε, κατάργησης της βίζας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και με τον Καναδά. Εάν είχαμε εγκρίνει αυτή την ε, πράξη λοιπόν θα ήταν αυτό αντιπαραγωγικό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας. Αγαπητή Μαριά, ο Καναδάς δεσμεύτηκε σε κοινή δήλωση, το γνωρίζετε αυτό, να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί μας για, με κατέθεση την πλήρη άρση των θεωρήσεων. Στις 11 Ιουλίου και στην Υπουργική δήλωση δεν μπορούσε να είναι πιο σαφής. Υποσχέθηκαν να επανέλθουν ε, το φθινόπωρο με μερμηνίες για την άρση των θεωρήσεων για την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ακόμα δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τις ημερομηνίε, όμως είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε καλά νέα από τον Καναδά συντόμως. Ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες μπορεί. Γιατί είπα, θα συνεχίσουμε την ίδια στρατηγική με την ίδια προσήλωση. Κυρία Χαλόμ, με τη ΣΥΠΑ, καμία από τις χώρες που δεν έχουν θεώρηση δεν ανταποκρίνονται στο 3% άρνηση των θεωρήσεων που ορίζεται στον Αμερικανική νομοθεσία. Το 2015 είχαμε ποσοστά απόρρεψης 3,5 για την Κύπρο, για την Πολωνία 6,4%, Βουλγαρία 17,3% και Ρουμανία 11,3% και Κροατία 5,3% απορρίψεις αιτήσεων. Το να δοθεί άρση της θεώρησης, να... κατάργηση μάλλον της θεώρησης, θα σήμαινε ότι η Αμερική θα έπρεπε να αλλάξει την νομοθεσία της και να ε, αλλάξει σημαντικά το κατόφλι του 3%. Καμιά όρεξη δεν έχει το Συμβούλιο, το Κογκρέσο, με συγχωρείτε, σαφώς να το κάνει αυτό. Αγαπητή Σεσίλια, δεν συμφωνώ μαζί σου. Κάναμε ένα σωρό πράγματα. Δεν με πιέζετε. Με πιέζετε, με και από κρυφά, αλλά εντάξει, μου αρέσει κιόλα η πίεση. Ε, τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν έχει δουλέψει για να εξασφαλίσει την ελεύθερη ε, μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών όσο γίνεται. Πριν τη διεύρυνση, του, διεύρυνση μάλλον του 2004 έφερε πολλές νέες περιπτώσεις μη αμοιβαιότητας. Ε, το 2005 18 κράτη-μέλη Σέγγεν είχαν απαιτήσει για βίζα από 8 τρίτες χώρες. Τώρα έχουμε 5 κρατημέλη και 2-3 χώρες με τις οποίες έχουμε ακόμα πρόβλημα. Η αμοιβαιότητα ανέκαθεν ήταν ε, προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε από αυτής μέχρι ότου να λυθούν όλες οι υποθέσεις μια αμοιβαιότητα, Ξέρω όμως ε, την ε, θέση σας. Βλέπετε, θέλω να κάνω μια πολιτική φύσης παρατήρηση. Ναι, έχουμε νομική ευθύνη. Φέρουμε νομική ευθύνη. Έχουμε και πολιτική ευθύνη έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίσουμε την άρση των θεωρήσεων για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και να μην αφήσουμε την καμία θεώρηση να ισχύει για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αλλά ξέρω ποιες είναι οι θέσεις σας, τις φωτίσατε, φωτίσατε το αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς και σας είμαι ευγνώμων και Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι, Κλοντ, που με καλέσατε και για αυτή την πορεία ξεκάθαρη, ειλικρινή και επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Και Ε, ξέρετε ότι πάντα τηρώ τι υποσχέσει μου στην Επιτροπή μου, γιατί σα θεωρώ δική μου οικογένεια, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα κρατήσω λοιπόν αυτή τη στάση σε όλε τι φάσει της και θέλω και πάλι να σα ευχαριστήσω που μου προσφέρατε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε, αλλά μια στιγμή. Αν δεν υπήρχε διαδικαστικό από τη Σόφη, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση καταλαβαίνω σωστά, μπορώ να συνοψίσω την απάντησή σας ότι λέτε ότι αρνούμε επίτροπος να φέρω σε πέρα στα καθήκοντά μου επειδή οι πολιτικές, τα πολιτικά επιχειρήματα υπερισχύουν των νομικών και άρα έτσι ε, τα δικαιώματα των πολιτών έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Έτσι συνοψίζεται η απάντησή σας σωστά. Αν ναι, τότε θα συμφωνήσω με τη συνάδελφο Βίλστρομ ότι μπορούμε να πάμε στο δικαστήριο εφόσον δεν φέρετε σε πέρα στα καθήκοντά σας. Πρόεδρος, ωραία. Ακούσαμε το διαδικαστικό. Εντάξει, δεν είχαμε φανταστεί ότι θα ήταν όντως διαδικαστικό. Μόνικα, τι, τι λες. Αν θέλετε. Εντάξει, είχαμε ένα μικρό επεισόδιο. Ο κύριος Διαθετεμέρα, ο συζητητής, δεν ξέρω, μήπως ο κύριε Διαθετεμέρα θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ο συζητητής, ναι, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ναι, κύριε Επίτροπε, πράγματι έχουμε μια πολιτική συζήτηση. Είπα όμως και πριν ότι πρόκειται για συζήτηση διαδικασίας επίσης και του κανονισμού 539. Αυτό που ακούσατε σημαίνει το εξής. Εμείς θα επιμείνουμε στις απαιτήσει μας. Θα είμαστε επίμονοι. Το λέω. Το είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Μωράης, το είπα και εγώ. Θα συμβιώσουμε με αυτήν την απέτηση και την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην υπάρχει παρεξήγηση γι' αυτό. Θα υπάρξει πίεση. Τώρα, το τι θα κάνει το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κάτι διαφορετικό από το τι θα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανεξάρτητο. Από πλευρά στρατηγικής σημασίας θα έλεγα ότι η στρατηγική συνήθως δεν δημοσιοποιείται, η στρατηγική ασκείται. Αλλά εγώ θα σας πω ποια είναι. Ξεκινήστε με την κατεξουσιοδότηση πράξη και δείτε πώς θα αντιδράσει το Κογκρέσο των Πολιτειών. Αλλά κάντε το. Προχωρήστε στην κατεξουσιοδότηση πράξη. Γιατί είναι το όπλο που έχετε, το εργαλείο σας για να προχωρήσετε σε επιτυχείς διαπραγματεύσεις. Και εκείνοι θα πρέπει κάτι να κάνουν, να αντιδράσουν, να κινηθούν. Μπορεί να πούνε, α, να το δουν σαν απειλή. Και να πούνε, α, τότε θα επιβάλλω και στους 28 την υποχρέωση θεώρησης. Ε, τότε όμως στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα υπάρξει συζήτηση Όπω θα υπάρξει συζήτηση όμως και με την κατεξουσιοδότηση πράξη, έτσι κι αλλιώ. Οπότε κάντε το και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν τελικά. Αυτοί θα πάρουν την απόφαση, εμείς και το Συμβούλιο. Κάντε το όμως, ξεκινήστε με την κατεξουσιοδότηση πράξη. Σε αυτό επιμένουμε. Και βέβαια καταλαβαίνουμε απόλυτα και δεχόμαστε απόλυτα αυτά που λέτε για την διπλωματική πίεση. Φυσικά είναι πολύ σημαντική μαζί με την πίεση που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρος. Ναι. Νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Μέρα. Θα ολοκλήρωνα με αυτό το διαδικαστικό εξής Είπα και πριν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινήστε τη διαδικασία. Αυτή είναι μια πολιτική πράξη στο κάτω-κάτω. Δεν μπορείτε εσείς να πείτε στη Λίμπε τι θα κάνει, να ε, την πατρονάρετε, εννοείται ποτέ. Αν κάνετε αυτό που λέει ο κύριος Δίαθ μέρα εδώ σας ε, βοηθάει, σας λέει ξεκινήστε τη διαδικασία και θα δείτε μετά τι θα γίνει. Αυτό σας ζητάμε λοιπόν. Μην έχετε καμία αμφιβολία για το τι επιθυμεί πραγματικά η Επιτροπή μας. Θα έχουμε την προφορική ερώτηση, θα έχουμε συζήτηση στην Ολομέλεια και θα τα ξανακούσετε συνεπώς από την Επιτροπή μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει και πολιτική διάσταση, αντιλαμβανόμαστε και τις υποχρεώσεις σας. Πάντως νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να τα πω καλύτερα από ό,τι τα είπε ο κύριος Ντιεθ και νομίζω ότι αυτή ήταν η καλή απάντηση σε αυτά που είπε και η κυρία Σόφι ότι υπάρχει υποχρέωση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει βέβαια και πολιτική διάσταση. Και έπειτα οι πολίτες των ενδιαφερόμενων χωρών καταλαβαίνετε ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν αρχίζει αυτή η διαδικασία για την κατεξοδότηση πράξη. Θέλετε να απαντήσετε παρακαλώ. Τους πολιτικούς ε, δεν πρέπει να τους βάζετε μπροστά σε ένα μικρόφωνο αν θέλετε να σας πούνε κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ θα κάνω μια κλίση. Πιέστε περισσότερο εμάς με επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ κύριε Επίτροπε. Colleagues, um, Συνάδελφοι, σημείο 11, αλλά είναι στο δρόμο ο εισηγητής για το σημείο 11 που είναι το επόμενο. Οπότε θα διακόψουμε για λίγα λεπτά. Λοιπόν, αν θέλετε να συμμετέχετε στη συζήτηση, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα για το σημείο 11, την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. Ο εισηγητής είναι ο Ζώζεφ Νάγκη. Να κάνω ίσως μια σύντομη εισήγηση. Εξετάζουμε τις τροπολογίες. Είναι η ετήσια έκθεση, συνάδελφοι, για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση. Όπως γνωρίζετε, είναι μία από τις βασικές ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής μας, καθώς περιλαμβάνει μία ε, λεπτομερή ανάλυση διαφόρων θεμάτων στην Ένωση. 986 τροπολογίες κατατέθηκαν φέτος για το σχέδιο έκθεσης και... Ο εισηγητής ζήτησε να γίνει ανταλλαγή απόψεων και θα του ζητήσω άμεσα να πάρει τον λόγο. Οπότε, παρακαλώ, ας αρχίσουμε την ανάλυση των 986 τροπολογιών. Είστε έτοιμος και εισηγητά. Μάλιστα, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Uh, ε, need Thank you for all colleagues. Uh, uh, Ευχαριστώ ε, όλους τους συναδέλφους που έστειλαν ε, τις ε, τροπολογίες τους για την έκθεση. Έχουμε 986 τροπολογίες μάλιστα και είναι κάτι παραπάνω από αρκετέ. Παίρνει κάποιο χρόνο αυτό με τη μετάφραση και τώρα προσπαθούμε να τις συνοψίσουμε σε συμβιβαστικές. Έχουμε 111 τροπολογίες μόνο για τα εκτιμώντας και 126 για τα, τις ε, αιτιολογικές σκέψεις. Φανταστείτε τι γίνεται λοιπόν. Προσπαθούμε να φτιάξουμε συμβαστικές γιατί δηλαδή θα περάσουμε μια μέρα ψηφίζοντας ε, την έκθεση αυτή. Τώρα, να σας πω πώς δουλεύουμε. Δεν παίρνουμε... Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν παίρνουμε τροπολογίες ε, για τα θέματα του 2016. Είναι αυτό πολύ σημαντικό γιατί πολλές τροπολογίες αφορούν θέματα του 2016. Ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε την έκθεση για το 2015, Ας πούμε, για το ψήφισμα για την εφαρμογή της οδηγίας για την, ε, για την εμπορία ανθρώπων. Έχουμε την ίδια οδηγία σε μια έκθεση, σε ένα σχέδιο έκθεσης. Ε, δεν παίρνουμε επίσης τροπολογίες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου κάνουν συστάσεις για όλες τις υποθέσεις που βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την επικάλυψη. Έχουμε τροπολογίες τώρα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου. Η κυρία Σόφη Ίντεβελτ κάνει σπουδαία δουλειά σε αυτή τη φάση για την έκθεσή μας και δεν ε, θέλουμε να όμως να αλλάξουμε τη δική της έκθεση, ούτε έχει νόημα να επικαλύπτουμε, να κάνουμε δύο φορές το ίδιο πράγμα με τις τροπολογίες και γι' αυτό και προσπαθούμε να δούμε την έκθεση από την οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές ε, τροπολογίες στάλθηκαν από την ε, από το Intergroup για τα παιδιά, για, το, για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Προσπαθούμε εμεί να μιλήσουμε για ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας των παιδιών με ένα σύστημα κυδαιμόνιας όπου τα κράτη-μέλη θα μοιράζονται τις πληροφορίες μεταξύ τους. Ε, θα υπάρχει και ένα νέο σύστημα, ένα νέο κεφάλαιο για τα ψηφιακά ε, δικαιώματα. Επίση πολύ σημαντικό θέμα και μιλάει για το πώς οι νέες τεχνολογίες συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως τα ντρόν ή τα, η επιγραμμική παρενόχληση, τα δικαιώματα των παιδιών στο ίντερνετ και εδώ λοιπόν καλύπτουμε πολλά θέματα Δεν θέλω να ε, διευρύνω τη συζήτηση για θέματα τα οποία είναι αντικείμενα μεμονωμένων εκθέσεων. Οπότε καταλάβετε παρακαλώ ότι πρόκειται για 986 τροπολογίε που δεν μπορούσαν όλες να ενταχθούν εδώ σε αυτή την έκθεση και με την πλήρη τους διατύπωση και πραγματικά κάνουμε πολύ σκληρή δουλειά προσπαθώντας να φτιάξουμε συμβιβαστικέ που να καλύπτουν όλες τις ιδέες που μας στέλνετε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε μια Ε, πλήρη εικόνα για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση το 2015. Ευχαριστώ, Ζώζη. Πολύ δύσκολη δουλειά, τόσες τροπολογίες. Ε, θέλουν διάφοροι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο για αυτές τις τροπολογίες ή Κριστίν. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποιε τροπολογίε που καταθέσαμε μαζί με τη συνάδελφο Σιβίκη Γιάννη, που στόχο έχουν να εμπλουτίσουν αυτήν την έκθεση και που δεν θεωρούμε πως είναι λεπτομέρειε ούτε αφορούν το 2016. Κατά προτεραιότητα θεωρήσαμε πως έπρεπε περισσότερο να διευκρινιστεί ε, το τι σημαίνει η βία κατά των γυναικών που είναι βασική παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά πρόκειται και μια βία η μορφή διάκρισης που είναι αίτιο και συνέπεια των ανισοτήτων ε, ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες. Αυτό το φαινόμενο αγγίζει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίκτυπο στα θύματα αλλά και στη κοινωνία ε, στο σύνολό τη. Είναι ε, αξιοθρύνητο ότι μια γυναίκα ή μια γυναίκα δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τη βία μέσα στην Ένωση στην οποία ζουν. Είναι πήγον λοιπόν να γίνουν πολιτικέ ευρωπαϊκέ για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών που ε, γίνεται που υπήρχε και το 2015. Πρώτον, η κύρωση της σύμβασης της ε, Κωνσταντινούπολης για την Ένωση αλλά και για τα κράτη-μέλη, η τα Κομισιόν θα πρέπει αυτό να το ξεπεράσει και να προτείνει ειδική οδηγία για το θέμα. Επιπλέον θέλουμε να επιμείνουμε για δύο συγκεκριμένα ε, σημεία, ότι καταρχάς πρέπει να, προστατευθούν όλα τα θύματα σεξιστικής βίας και τα άτομα ε, LGBT, γιατί κάτι τέτοιο είναι αδικαιολόγητο σε κάθε περίπτωση. Επίσης με τις οπολογίες μας τονίζουμε ότι τα μέτρα καταπολέμησης της εμπορίας των ανθρώπων δεν θα πρέπει να πλήττουν τα δικαιώματα των θυμάτων της εμπορίας, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ε, μνήμα για τους ε, ασυνόδευτους ανήλικους. Επίσης θα πρέπει η Ένωση να υπογράψει την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων. Κάτι ακόμα σημαντικό που δεν είναι στην έκθεση αλλά που αφορά την προστασία του κράτους δικαίου. Είναι μια βασική αρχή επί της οποίας οικοδομήθηκε η Ένωση. Ε, και το 2015 ήδη ήταν επίκαιρο αυτό το θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρήσαμε πως ήταν απαραίτητο να στηρίξουμε το κράτος δικαίου, ναι, με την έκθεση της ε, Σοφία Ίντερβελ ναι, το 2016, αλλά έπρεπε ήδη να το συμπούμε και για το 2015, ώστε τα κράτη μας να στηρίζουν το κράτος δικαίου καθημερινά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Άννα Μαρία Κοράτσα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Γιώζεφ Νάγκη ε, επειδή συμπεριέλαβε τόσα πολλά και τόσο σωστά στις τροπολογίες ε, για το κεφάλαιο για τα δικαιώματα των παιδιών. Εγώ είμαι συμπρόεδρος ε, του Intergroup για τα δικαιώματα των παιδιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω οι συνάδελφοι να το στηρίξουν αφορά εκεί, την συμπερίληψη της ε, προστασίας των παιδιών ε, online επιγραμμικά, να απογορεύεται το profiling, το φακέλωμα, αλλά και η άμεση διαφήμιση προς τα παιδιά, η βία κατά των παιδιών και ελπίζω πως θα μπορέσετε όλοι σας να το στηρίξετε. Ε, Εφόσον πρόκειται για, δε, για έκθεση για τα ανθρώπινα, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα με την άνοδο της άκρα δεξιά θα πρέπει να θυμίσουμε ακόμη μια φορά ότι ομοφοβία, η οχλαγωγία, η ε, ε, ελευθερία σεξουαλικής προτίμησης είναι θεμελιώδη δικαιώματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να θυμίσω ακόμα μια φορά στο Συμβούλιο και σε όλους ότι η διοδηγία κατά των διακρίσεων που έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει. Πρόκειται για θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελπίζω πως η εκθέση αυτή θα είναι μια ευκαιρία ώστε να προχωρήσουμε στα θέματα, αφορούν, ε, στα θέματα κατά των διακρίσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Κινίτσι. Τσινίτσι. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Νάγκη και όλους τους συζητητές για την τεράστια δουλειά τους, αλλά και κυρίως για τα όσα θα κάνουν στη συνέχεια. Θέλω να τον ευχαριστήσω που έδωσε μεγάλη προσοχή και εγώ συμφωνώ με την έκκληση της συναδέλφου Κοράτσα Μπίλτε ως ε, ε, συμπροέδρος της ομάδας για τα παιδιά ε, και θέλω να μιλήσω για την ανάγκη να μπουν μέσα στα θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία του παιδιού σε σχέση με τους κινδύνους ε, που προέρχονται από το διαδίκτυο και αναφέρομαι κυρίως στη δυνατότητα να, εντάξει, να, να, να, στηριχθεί το δικαίωμα στη λύθη, δηλαδή να μπορεί να, να, να αφαιρείται ε, περιεχόμενο το οποίο είναι προσβλητικό ή αναξιοπρεπέ. Αυτό έχει οδηγήσει δυστυχώ και στη χώρα μου σε ε, αυτοκτονίε. Αυτό επηρεάζει κυρίω τι γυναίκε αλλά και του ανήλικου, ανήλικους οι οποίοι πολύ συχνά δι, ε, πέφτουν θύματα του κυβερνομπούλινγκ ε, και θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον συναδελφό άλλη μια φορά για την σπουδαία του δουλειά και θα πρέπει και αυτές οι μορφές προστασίας να ε, ενταχθούν ε, στις, ε, στο κείμενο. Κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρους που δεν μπορεί να είναι εδώ, που είναι σκιώδης εισηγητής και ζητά συγγνώμη γι' αυτό. Το διαβάζω, λέει η κυρία Κάφμαν. Λέει, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές που δούλεψαν πάνω στις τροπολογίες, που είναι πολλές και φέτος. Μπορώ να πω ότι οι τροπολογίες μας έχουν σαν στόχο να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής και να συμπεριλάβουν περισσότερες ομάδες και περισσότερες κατηγορίες που λείπουν. Θέλω να αναφέρω επίσης το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου είναι προϋπόθεση για να τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως έχουμε ακούσει και από την Επιτροπή. Πολλά θέματα μας ε, κάνουν να πιστεύουμε ότι υπήρχαν πολλές ε, παραβιάσεις στην Πολωνία, για παράδειγμα, οπότε είναι δύσκολο να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή για τα θεμελιώδη δικαιώματα χωρίς να αναφέρουμε αυτά τα ζητήματα και να προτείνουμε λύσεις. Βέβαια δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τις παραγράφους, αλλά αν μη τι άλλο στις τροπολογίες μας να αντικατοπτρίζονται. Πιστεύουμε ότι τα δικαιώματα των ΛΟΕΔ λείπουν συστηματικά από τέτοιες εκθέσεις, γι' αυτό και εμείς έχουμε υποβάλει διάφορες τέτοιες τροπολογίες. Όσον αφορά τώρα την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, επίσης υπάρχουν πολλά ζητήματα το θέμα της ε, βίας σε βάρος ε, των ε, γυναικών είναι κάτι που έχει να κάνει με την ζώτα των δύο φίλων. Θα πρέπει να, να υπογραμμίσουμε περισσότερο επίσης τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, κυρίως μετά από τα πρόσφατα γεγονότα στην Πολωνία και την ομοθεσία για την άμβλωση που ισχύει στην Πολωνία και την Ιρλανδία. Όσον αφορά τους Ρώμα, διαγράφουμε την παράγραφο για τα παιδιά αυτά γιατί ε, μιλάει συγκεκριμένα για τους Ρώμα και παρουσιάζει πολύ απλοποιημένη εικόνα των ανθρώπων αυτών που δεν είναι σωστή. Στην Ουγγαρία είδαμε ότι άστεγοι μερικές φορές θεωρούνται εγκληματίες, ε, καταδικάζονται ε, συστηματικά με αποτέλεσμα η δερματοποίηση να διονύζεται. Η ελευθερία έκφρασης επίσης συνείδησης και θρησκείας. Πρέπει να προστατευτεί η ελευθερία του τύπου και των δημοσιογράφων. Πρόσφατα έκλεισε η ημερήσια εφημερίδα στην Ουγγαρία μετά από πολιτικές παρεμβάσεις στον πλουραλισμό του τύπου. Θέλουμε λοιπόν εγγύησει, όπως επίσης και για τη θρησκευτική ελευθερία, να λάβουμε επίσημας, επίσης ε, υπόψη μας τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος ε, ορισμένων ομάδων, αντισημιτισμός κτλ. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι είμαι υπέρ επικοδομητικής συζήτησης, να δεχτώ συμβιβασμούς, αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς προκειμένου να μπορούμε να εγκρίνουμε στην Επιτροπή μας την έκθεση αυτή τον αύριο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κανένα άλλος? Όχι. Ωραία. Ο εισηγητής πάλι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και σας ευχαριστώ Όντως, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και η δουλειά θα είναι σκληρή με τους σκιώδες εισηγητές προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις απόψεις. Ευχαριστώ πάντως για τις τροπολογίες που υποβάλλατε. Κυρίως για τα δικαιώματα των παιδιών. Είμαστε στην αρχή της δουλειάς και είπα ήδη ότι θέλω να επικεντρωθώ σε κάποια ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται συχνά από άλλες εκθέσεις. Είναι καλό λοιπόν να συμπεριλάβουμε ό,τι αφορά το 2015 για αυτά. Τα δικαιώματα των παιδιών σε όλα τα κεφάλαια επικεντρωνόμαστε στα παιδιά. Θέλω να αντιδράσω στο εξής. Κράτος δικαίου. Δεν θέλαμε να καταλήξουμε στο blaming and shaming, να καταδεικνύουμε δηλαδή ποιος και να κατονομάζουμε δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να το θέλουν για λόγους εθνικής πολιτικής, αλλά δεν είμαστε σε άλλο επίπεδο και πρέπει να λέμε γενικά τα πράγματα. Τώρα για τους ζητιάνους, τα παιδιά ζητιάνους. Νομίζω ότι υπάρχει παρεξήγηση. Εδώ δεν κατονομάζουμε τους Ρώμα. Πρέπει να το συζητήσουμε όμως. Γιατί ακόμη και σε αυτή την πόλη, σε όλες τις πόλεις, δεν έχει να κάνει με την ε, εθνότητα την καταγωγή των παιδιών, όταν μιλάμε για δικαιώματα των παιδιών δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια επειδή ίσως ενοχληθεί ε, η μία ή άλλη εθνότητα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και προσβλέπω στην καλή συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστούμε. 17 Νοεμβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία. Τώρα, ψηφοφορία 10.40. Ε, μέχρι τις 10.40 λοιπόν θα διακόψουμε. Να είσαστε εδώ όμως ακριβώς. Α, έχεις διαδικαστικό. Παρακαλώ. Ναι, ναι, διαδικαστικό. Ίσως να συζητήσουμε τώρα για τον τριμερή διάλογο όσον αφορά τον κώδικα θεώρησης γιατί κάποιες χιλιάδες πρέπει να πάμε σε άλλες συνεδριάσεις. Η κυρία Βαλέρο, για παράδειγμα, πρέπει να πάει σε κάποια άλλη συνεδρίαση αργότερα, ενώ θα ήθελε να συμμετάσχει στη συζήτηση αυτή για την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά τον κώδικα θεωρήσεων. Πρόεδρος, αν συμφωνούν όλοι, δεν έχω αντίρρηση. Και ευχαριστώ, Φερνάντο. Ωραία, ε, όσοι θέλανε καφέ, χάσανε. Κι εγώ ήθελα, ήθελα διάλειμμα, το ομολογώ, λέει ο πρόεδρος, αλλά θα κάνω τη δουλειά μου. Και θα πάμε στο θέμα αυτό της αναδιατύπωσης θεωρήσεων. Σημείο 4 λοιπόν. Πρόκειται για την παρουσίαση τον Μάρτιο ήδη για τον ενωσιακό κώδικα θεωρήσεων. Αναδιατύπωση έγιναν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και με την Ολλανδική Προεδρία ξεκίνησαν. Ε, αλλά βέβαια τώρα είμαστε στην ε, Σλοβακική Προεδρία. Όποιος θέλει το λόγο, ευχαρίστως. Εσύ, Φερνάντο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Ευχαριστώ όλους του συναδέρφους που μου επέτρεψαν να κάνω αυτήν την σύντομη παρουσίαση. Είναι μια σημαντική υπόθεση και έχουμε μια καλή ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τον κώδικα αυτό βάσει των άρθρων που προβλέπονται στη συνθήκη της Λισαβόνας για την ελεύθερη κυκλοφορία κλπ. Πρέπει να έχουμε μια κοινή πολιτική θεωρήσεων. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό κώδικα θεωρήσεων, όπως θα έπρεπε να είχαμε, και κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων που έρχονται από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, μετά την πρωτοβουλία της Επιτροπής, κολλήσαμε. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση στο Συμβούλιο. Προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση που να οδηγήσει σε συμβιβασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει με εμά, δηλαδή, με την Επιτροπή μας, ΛΥΜΠΕ. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη πολιτικής βούλησης για συμβασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορες σοβαρές συζητήσεις που έχουμε κάνει με το Συμβούλιο, ιδιαίτερα στους τριμερείς διαλόγους που είχαμε μέχρι τώρα. Ακόμα και χτες Είχαμε συνάντηση με τη Σλοβακική Προεδρία, με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μάτιους Ρούτ από τη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής ήταν εκεί για ολόκληρο το φάκελο. Εμείς δώσαμε σημασία στο θέμα των θεωρήσεων για θρεπιστικούς λόγους. Μετά συζητήσαμε τις γενικές διευκολύνσεις και τη συνεργασία με χώρες οι οποίες πραγματικά επιθυμούν να συμφωνήσουν με την επανεισδοχή από τις χώρες μέλη. Στη συνέχεια συζητήσαμε για τις κατεξουσιδότηση και τις εφαρμοστικές πράξεις, ε, οδηγίες, εφαρμογή κλπ. Και μετά έγινε παρουσίαση, ε, ορισμοί για τις διευκολύνσεις που προτείνονται Τέλος, για τον μηχανισμό θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων. Ε, λοιπόν, σε κανένα από αυτά τα κεφάλαια δεν είδαμε κάποιο σημάδι ότι υπάρχει βούληση από το Συμβούλιο να μετακινηθεί προς τις δικές μας θέσεις. Εμείς δείξαμε ότι θέλουμε συμβασμό. Δείξαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι από την αρχική μας θέση του εισηγητή και των σχεδόν εισηγητών να μετακινηθούμε προς το Συμβούλιο. Από τη θέση της ΛΥΜΠΕ λοιπόν, εμείς μετακινηθήκαμε προς τη δική τους κατεύθυνση. Όμως από τη δικιά τους την πλευρά δεν πήραμε κανένα σημάδι μετακίνησης προς τη δικιά μας θέση. Και αν ήταν η μόνη φορά Εντάξει, αλλά δεν είναι. Σε πάρα πολλούς φακέλους ε, καθυστερούν, ε, ε, χασομεράνε και παρακολύουν τελικά τη διαδικασία. Αρνούνται να κατανοήσουν ότι είμαστε συνομοθέτες κι εμείς. Νομίζουν ότι είναι μόνοι τους που με συμφωνίες πλαίσιο θα προχωράνε. Αυτό ήταν κάποτε. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας γίναμε συνομοθέτες. Άρα είμαστε ουσιαστικοί προκειμένου να προχωρήσει η νομοθεσία. Δεν προχωράει όμως, γιατί εκείνοι δεν μετακινούνται. Και θέλω να προσθέσω εδώ απλώς, για να καταλάβετε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, ότι εδώ δεν πρόκειται για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Εμείς, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητάμε τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Και γιατί, γιατί είχαμε διάφορες ακροάσεις με νομικούς, με ανθρωπιστικές οργανώσεις, με κυβερνητικές οργανώσεις, εκκλησίες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, που εκφράζουν ανησυχίες για την τραγική κατάσταση από την ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη που ονομάζουμε προσφυγική. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις που δεν θέλουν έτσι κι αλλιώς να μετακινηθούν. Όχι. Δεν θέλουν να συμβιβαστούν ούτε για τις διευκολύνσεις, ούτε για τη συνεργασία, ούτε για την επανεισδοχή, ούτε για τις κατεξουσιοδότηση και τις εφαρμοστικές ε, πράξεις. Ε, τίποτα, ακόμα και αυτά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο θέμα των θεωρήσεων. Ή για τους ορισμούς, ποιοι είναι οι στενοί συγκινείς, και για το θέμα των πολλαπλών ε, εισόδων, των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνουν ότι για να προχωρήσει αυτή η νομοθεσία χρειάζονται τη δικιά μας συναπόφαση. Χρειάζονται τη δικιά μας εμπλοκή στην νομοθετική διαδικασία. Αν αυτό δεν το καταλάβουν, και σας λέω όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε πολλούς σημαντικούς ε, φακέλους για το άσυλο, για την αναθεώρηση του Σέγγεν, και πολλούς άλλους, δεν θα υπάρξει καμία νομοθετική πρόοδος όσο δεν μετακινείται το Συμβούλιο. Στο τέλος της θητείας θα είναι καταστροφική η κατάσταση. Αυτό πρέπει να τους ανησυχήσει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη αποτυχάνει. Και αυτά σας τα πάρα πολύ σοβαρά. Ε, ένας ε, σκιώδης εισηγητής, η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ βρίσκομαι. Αυτά που είπε ο Χαν Φερνάντο απηχούν και τι δικέ μου απόψει. Δεν έχουμε ακόμη ανταπόκριση από το Συμβούλιο Υπουργών και δεν είναι μοναδική περίπτωση. Τα ίδια βλέπουμε και στον τριμηρή διάλογο για τον μηχανισμό αναστολή, όπου αυτοί του Συμβουλίου δεν κάνουν καμία κίνηση. Η δε απάντηση που λάβαμε για την ανθρωπιστική βίζα ήταν «Μα έχουμε ούτως ή άλλως τις εθνικές βίζες, να χρησιμοποιήσετε αυτές». Μα αυτά δεν αποδίδουν, δεν λειτουργούν. Και όταν γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργούν και ότι καμιά χώρα δεν τις χρησιμοποιεί, τότε πρέπει να κάνουμε κάτι και να επιφέρουμε κάποια αλλαγή. Πλήρη υποστήριξη λοιπόν προς τον εισηγητή μας και σε τριμερείς διαλόγους κλπ. Είναι σημαντικό να είμαστε, να φανούμε ισχυροί, διότι το Συμβούλιο θα προτιμούσε να είμαστε εμεί κάπου αλλού και να μην βγαίνουμε ούτε καν να προτείνουμε πράγματα. Όμω είμαστε συνομοθέτε και αυτό οφείλει να το κατανοήσει το Συμβούλιο. Αυτά είχα μόνο να προσθέσω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Το Λαϊκό Κόμμα, κύριο Μπέκερ. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Σημειώνω αυτά που έχω ήδη άλλωστε πει κατά επανάληψη και σε προσωπικές συνομιλίες, ότι μέχρι σήμερα καμία παρέμβαση Καμία παρέμβαση δεν έχω κάνει στην προσωπική διεύθυνση των συζητήσεων του διμερού διαλόγου από τον εισηγητή. Αυτό το θεωρώ αυτονόητο, διότι οφείλει κανεί να είναι πιστό στην απόφαση τη Επιτροπή, τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή δηλαδή. Θεωρώ όμω ότι η κατάσταση όπω διαμορφώνεται στον τριμερή διάλογο είναι διαφορετική από αυτήν που εξηγεί ο εισηγητής. Ναι μεν αντιλαμβάνομαι ότι το Συμβούλιο δεν δείχνει μεγάλη διάθεση να προωθήσει την ανθρωπιστική βίζα με την μορφή που περιλαμβάνεται στην ε, τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Αυτό όμως είναι φυσικό, διότι το Συμβούλιο με το δίκαιο του προβάλλει το επιχείρημα, άλλωστε το έχουμε πει και εμείς, αλλά δεν το ξανακάναμε, ξανακάναμε θέμα στον τριμή διάλογο τώρα. Λέει λοιπόν ότι η ρύθμιση της ανθρωπιστικής βίζας δεν εμπίπτει στις νέες ρυθμίσεις του κώδικα θεωρήσεων που έχει να κάνει με επιχειρηματίες, τουρίστες και καλλιτέχνες. Και αυτό είναι το μοναδικό σημείο όπου ασκεί αντίσταση το Συμβούλιο σε όλα τα άλλα θέματα δεν βλέπω αρνητική στάση, βλέπω μάλλον μια διαπραγματευτική τακτική η οποία έχει κάποια λογική. Και όποιος έχει διεξαγάγει διαπραγματεύσεις μέσα στα πλαίσια τριμερών διαλόγων, την αντιλαμβάνεται ως συνήθι διαπραγματευτική τακτική. Δηλαδή, δεν προχωρούν σε ένα συμβασμό εφόσον θέλουν να συμβαστούν σε κάποια σημεία κεντρικής σημασίας. Εγώ θεωρώ ότι τελικώ ο συμβασμό θα είναι δυνατόν. Για το θέμα των στενών συγγενών, νομίζω πρόκειται για μια διάσταση όπου είναι, υπάρχουν οι ορισμοί μέσα στα θεμελιώδη δικαιώματα του καταστατικού χάρτη της Ένωσης. Στενοί συγγενείς δεν είναι οι παππούδες και τα εγγόνια. Και εγώ είμαι κατά της άποψης να σταματήσει η περαιτέρω συζήτηση στον τριμήρη διάλογο. Αυτά που ζητεί ο εισηγητής από το Συμβούλιο, δηλαδή ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της ανθρωπιστικής βίζας, αυτό το έχει λάβει. Και αυτό μπορεί να συμφωνηθεί εύκολα εφόσον και τα τρία θεσμικά όργανα λάβουν την υποχρέωση στην επόμενη νομικοτεχνική επεξεργασία του resettlement να περιλάβουν στη ρύθμιση και την ανθρωπιστική βίζα, όπως εμείς την έχουμε άλλωστε περιλάβει στον συμβασμό. Να μην χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την ρύθμιση του Visa Code, στρέφοντάς την τελικά κατά εκείνων για τους οποίους έχει φτιαχτεί. Δηλαδή σημαντικούς και για την Ευρώπη. Επιχειρηματίες από τρίτες χώρες, τουρίστες, περιηγητές, ταξιδιώτες από τρίτε χώρε και καλλιτέχνε. Να μην βάλουμε εμεί εμπόδια μόνο επειδή το Συμβούλιο, το αναγνωρίζω αυτό, τακτικά εμφανίζεται αδέξιο, α το πω έτσι. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ο εισηγητή σε πολλές φάσεις της διαπραγματεύσεω δείχνει μια πραγματικά, πραγματική δεξιότητα και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει εν τέλει αλλά να μην υπαναχωρήσουμε εμείς τώρα σε μια ε, στάση που να δείχνει ότι μόνο εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Η Σεσίλια Βίκστρομ. Θα είμαι σύντομη διότι ο δικός μας και ο Δεπρέ Ντεπρέ δεν είναι παρόν και με παρακάλεσε να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι στηρίζει τον εισηγητή απολύτως, συμπαρατάσσεται μαζί του και ελπίζει ότι θα προκύψει ένα θετικό αποτέλεσμα. Με την ευκαιρία θα ήθελα να μεταφέρω το ίδιο μήνυμα και σε ό,τι αφορά την έκθεση Guillaume για την ασφαλή χώρα προέλευσης. Και εκεί λοιπόν ο δικός μας σκιοδησηγητής στηρίζει την ε, προσπάθεια της κυρίας Guillaume. Ευχαριστώ. Επειδή αλλάξαμε την σειρά, δεν θα έχουμε Προεδρία και Επιτροπή εδώ. Θα επανέλθουμε όμως Ευχαριστώ, Χουάν Φερνάντο, που ε, πρότεινε να συζητήσουμε το θέμα τώρα. Ίσως έχουμε και ε, την αναφορά τώρα στον τριμήριο διάλογο από την κυρία Γκυγιώμα, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε στα λίγα λεπτά που μένουν. Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί. Τώρα δεν λειτουργεί ούτε του Πρόεδρου, δεν το έχει ανοιχτά ο Πρόεδρος, δεν ακούμε τίποτα. Δεν ακούμε τίποτα, ούτε από τον Πρόεδρο, ούτε τίποτα από την αίθουσα. Τώρα εντάξει, τώρα ακούγεται. Τώρα ακούγεται. Πρόεδρε, έλεγα ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε. Αν θέλετε να πάρω το λόγο, να πάρω το λόγο. Ό,τι θέλετε. Uh, Σε ένα λεπτό είναι η ψηφοφορία, οπότε θα αναγκαστούμε να περιμένουμε. Λοιπόν, για να μην έχετε την απορία αν δεν καταλάβατε, προσπαθούσαμε να συνοηθούμε αν θα έχουμε άλλο ένα σημείο πριν την ψηφοφορία επειδή είχαμε λίγο χρόνο πριν τις ψηφοφορίες, αλλά όχι αρκετό από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Αργότερα θα περάσουμε στην έκθεση Γκυγιόμ ή τέλο στην ε, παρουσίαση της κυρίας Γκυγιόμ. So colleagues, as soon as everyone has taken their seat, we'll begin the Καθίστε παρακαλώ όλοι για να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Σύντομα έχουμε δύο και έγκριση του χρονοδιαγράμματος. Όταν είσαστε έτοιμοι, αρχίζουμε. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Καλώς. Εσύ, Τόμας, το ξέρω ότι είσαι έτοιμος. Οι άλλοι δεν ξέρω. Αν είσαστε όλοι έτοιμοι, ας αρχίσουμε. Έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία σημείο 12 αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA στη Δανία. Ωραία, περιμένω λίγο ακόμα. Συνάδελφοι, σταματήστε τη συντονίστρια του ΕΛΚ να βάλει την κάρτα της. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου δεν τις ακούμε. Επόμενο, αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Καλώς. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Το σημείο 14 τώρα, που είναι η έγκριση του ετήσιου χρονοδιαγράμματος συνεδριάσεων της ΛΥΜΠΕ για το έτος 2007. Το έχετε το χρονοδιάγραμμα, έτσι, το εγκρίνετε. Καλώς, ευχαριστώ. Ωραία, τελειώσαμε με την ψηφοφορία και ευχαριστώ πολύ. Σημείο 15 τώρα. Αν δεν σκοπεύετε να μείνετε για να παρακολουθήσετε, τότε σας παρακαλώ αποχωρήστε ησύχως. Για το 15, δυστυχώς δεν έχουμε την εισηγήτρια, την κυρία Γκόμες, μάλλον θα είναι στο δρόμο. Θα έρχεται, οπότε τι να κάνουμε. Α, κυρία Γκυγιόμ, να, τώρα. Τι λέτε. Ωραία. Σημείο 3 λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι τώρα που είναι ο τριμερής διάλογος. Θα μας αναφέρει η κυρία Γκυγιόμ το τι έχει γίνει στον ε, διάλογο αυτό. Πρόκειται για θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγή για του σκοπού κοινών διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων στον τριμερή διάλογο. 13 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρο πρώτος τριμερής ε, διάλογος και η κυρία Γκυγιόμ θα μας ενημερώσει σχετικά. Παρακαλώ κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το πατήχαμε ένα πρώτο τριμερή διάλογο στις 13 Σεπτεμβρίου και ο επόμενος προβλέπεται στις 19 Οκτωβρίου. Έχουμε υιοθετήσει θέση εδώ στη Λίμπε, σας θυμίζω, στις 13, μάλλον διορθώνω μιλήτρια, στις 7 Ιουλίου που μας πέρασε. Το κείμενο είναι ποιότητας, πιστεύω. Ενισχύει την άποψη για εναρμόνιση Αναφέρεται στη μεθοδολογία επίσης όσον αφορά την αξιολόγηση των τρίτων χωρών και μιλάει και για έναν μηχανισμό προκειμένου η διαδικασία να προχωράει πιο ήπια και πιο γρήγορα. Έχουμε προβλέψει και ένα διαδικαστικό πλαίσιο επίσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουμε ενισχύσει. Οι συζητήσεις άρχισαν λοιπόν με το Συμβούλιο. Περίτω να σας πω για το πλαίσιο, αλλά στο πούμε καλύτερα, ότι οι συζητήσεις δεν θα είναι εύκολες για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο κατάλογος των χωρών που προτείνεται δεν έχει αξιολογηθεί κατά περίπτωση και δημιουργείται πολλές φορές ε, σύγχυση εξαιτίας των ενιών της ασφαλούς χώρας που νομίσαμε ότι θα διευθετούσε το προσφυγικό, πράγμα που δεν έγινε. Έπειτα νομοθετικά υπάρχει λίγο πρόβλημα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίμενε ότι θα προχωρήσουμε και για το άσυλο, αλλά επαναλαμβάνω ότι ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, που είναι το 2013, δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα. Που σημαίνει ότι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστια και όσον αφορά το περιεχόμενο και όσον αφορά την ε, διαδικασία βάσει της οποίας εργαζόμαστε. Έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά συντονισμού μεταξύ μας για να υπάρχει συνοχή στο αποτέλεσμα. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η έννοια του Ευρωπαϊκού Καταλόγου με ε, χώρες καταγωγής ασφαλής είναι κάτι που βλέπουμε σε όλα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που βρίσκονται προς διαπραγμάτευση. Εννοείται ότι συζήτησα και με τη Λάουρα Φεράρα, τη συνάδελφο, όταν μιλάμε για κανονισμό, διότι οι διατάξεις που προβλέπονται στον ευρωπαϊκό κανονισμό πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στον κανονισμό για τη διαδικασία που θα εγκριθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να σεβαστούμε τις ε, μέχρι τώρα θέσεις. Τώρα για το περιεχόμενο και την πρώτη συζήτηση τριμερούς διαλόγου, αλλά και τη συνέχεια. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, αλλά κινδυνεύουμε να κολλήσουμε με το Συμβούλιο σε πολλά σημεία. Για το θέμα της αναρμόνισης πρώτα απ' όλα. Γιατί εμείς αφαιρούμε τελικά, λέμε δηλαδή να μην υπάρχουν εθνικοί τέτοιοι κατάλογοι, αλλά ένας ευρωπαϊκός. Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί και όχι απλώς δεν συμφωνεί, είναι σαφώς κατά. Θέλει να συνεπάρχουν. Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Τρίτων Ασφαλών Χωρών, Ευρωπαϊκός, λοιπόν με τους εθνικούς, ενώ εμείς θέλουμε εναρμόνιση. Μάλιστα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη διάσταση απόψεων μεταξύ μας. το άλλο που συζητάμε είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όπως έλεγα και πριν, ενισχύσαμε κάποια δικαιώματα μέσω της άρσης προσφυγών και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στους ανήλικους και σε άλλες κατηγορίες και κυρίως στους ανήλικους τους ασυνόδευτους. Αλλά και εδώ, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ δύσκολο να δούμε τον ευρωπαϊκό κατάλογο εντελώς απομονωμένα. Και το άλλο περίπλοκο σημείο, το μεθοδολογικό. Εμείς θέλαμε να δώσουμε ειδικό ρόλο σε διάφορες οργανώσεις, για παράδειγμα την ΥΠΑ, Αρμοστία του ΟΗΕ ή σε άλλες μη κυβερνητικές διεθνείς οργανώσεις. Δεν λέω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, αλλά αν μη τι άλλο να χρησιμοποιήσουμε την πραγματογνωμοσύνη όλων αυτών για να βοηθηθούμε στη συνέχεια. Υπάρχει τώρα μια στρατηγική που δημιουργείται, γιατί φαίνεται ότι το Συμβούλιο για να παρακάμψει αυτά τα εμπόδια θέλει αναβολή. Και ενδεχομένως να δούμε το θέμα του καταλόγου αυτού μέσα στο φάκελο το διαδικαστικό. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Επίσης, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προχωρήσουμε γρήγορα στην έγκριση. Ειλικρινά η συζήτηση με τους σκιώδεις ήταν βέβαια σύντομη. Αλλά ήδη και φαίνεται και από τη θέση του Ντεπρέ, κανείς δεν θέλει ο ίδιος να έχει την καυτή πατάτα. Όλοι θέλουν να το κλειτώσουν αυτό, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο όσο δεν διακανονίζεται ποιε είναι ασφαλείς χώρε και ποιε όχι. Και έπειτα στρατηγική αυτή το άλλο που δεν είναι ικανοποιητικό είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα που ενισχύουν τη θέση του Κοινοβουλίου για τον ε, κατάλογο αυτό. Αν από το κείμενο τα βγάλουμε όλα αυτά, τότε ο κατάλογος στον οποίο, μάλλον ο κανονισμός στον οποίο θα καταλήξουμε, θα έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, Πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις, θα είναι δύσκολες, αλλά το ξέρουμε, και πρέπει να επιμείνουμε στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πλήρης η ανάπτυξη του θέματος. Δεν ξέρω αν κανείς επιθυμεί να λάβει το λόγο. Αν όχι, σας ευχαριστώ και πάλι Σιλβί. Και πρόκειται βεβαίω για, πολύ για σημαντικό θέμα τη δέσμη αυτή. Ακόμη δεν έχει έρθει η κυρία Γκόμε. Ευχαριστώ λοιπόν, ε, Σιλβί. Η κυρία Γκόμε ακόμα δεν είναι παρούσα, άρα δεν μπορούμε να έρθουμε στο θέμα υπαριθμού 15. Να δούμε αν ίσως μπορούμε να έρθουμε στο 5. η ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ενώσεως κατά των απατών. Η κυρία Κινίτσι είναι παρούσα. Δέχεστε να παρουσιάσετε το θέμα και θα δούμε είναι και οι άλλοι αρμόδιοι παρόντες. Συμφωνείτε, συνάδελφοι, αλλάζω βεβαίως διαρκώς την ημερησία διάταξη, αλλά αναγκάζομαι να το πράξω αυτό λόγω των απουσιών. Η κυρία Χόλμαϊρ, μία ερώτηση, διότι η κυρία Τσινίτσι αύριο δεν μπορεί να είναι παρούσα αν έχουμε χρόνο μπορούμε να συζητήσουμε την τρομοκρατία σήμερα, αν λείπουν και άλλοι συνάδελφοι, διότι θα κάνουμε ένα σύντομο state of play και μετά μπορεί και η κυρία Κινίτσι που είναι σήμερα παρούσα να συμμετάσχει και αυτή, εάν βεβαίως είναι δυνατόν αυτό. Καλή ιδέα και πάλι βεβαίω υπό την αίρεση ότι μου δίνει την άδεια η Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Ευχαριστώ λοιπόν που ε, είστε τόσο ευέλικτοι Θα θέλατε, ε, Κατερίνα, να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ναι, μπορούμε να αρχίσουμε. Μάλιστα, τέλεια. Ευχαριστώ, Κλοντ, και ευχαριστώ και τη Μόνικα, γιατί όντως μπορέσαμε μαζί να δούμε αυτή την οδηγία κατά της ε, τρομοκρατίας. Όσον αφορά τώρα τη γνωμοδότηση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ε, για την οποία είμαι συγγήτρια, σήμερα συζητάμε για αυτό το θέμα προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και καταπολέμηση των απατών, αλλά τη απουσία της ετήσιας έκθεσης, ε, την οποία αναμένουμε για την αρχή του χρόνου και άρα στην πράξη, δεν γνω... και στην πράξη όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα δημοσιευθεί. Ε, θα είχαμε έτσι πληρέστερο πλαίσιο ε, και θα μπορούσαμε να έχουμε καταλάβει καλύτερα πώς προχωράει αυτό το φαινόμενο, πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο για να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα αλλά και για να συνειδητοποιήσουμε τον αντίκτυπο των μέτρων που έχουν ήδη ε, ληφθεί. Ε, το σίγουρο είναι ότι απάτες συνεχίζουν να γίνονται και ότι είναι διαδεδομένα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, και μάλιστα οι απώλειες ανέρχονται σε 5 ε, δισεκατομμύρια το χρόνο και έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Είδαμε με τον καιρό να πολλαπλασιάζονται τα νομοθετικά κείμενα και να γίνονται διάφορες προσπάθειες, όμως σίγουρα έτσι φαίνεται πως υπάρχει η ανάγκη για προστασία σε επίπεδο της Ένωσης και όχι μόνο σε επίπεδο των μεμονωμένων χωρών, και επιβεβαιώνεται ωστόσο ότι το φαινόμενο συνεχίζει να υπάρχει και άρα είναι απαραίτητο να υπάρξει παρέμβαση για να προστατευθούν ε, οι πολίτες αλλά και για να παρακολουθείτε και η κατάσταση και να δίνουμε και λογαριασμό στους πολίτες για την ορθότητα των ευρωπαϊκών λογαριασμών. Γνωρίζουμε εξάλλου ότι ότι να πάτε εύκολα κανείς περνάει και στη διαφθορά και ότι μέσω της διαφθοράς χρηματοδοτείται και το οργανωμένο έγκλημα και όπως γνωρίζουμε και η δρομοκρατία. Πρόκειται για παραπομπές οι οποίες εξυπηρετούν το να, το να υπογραμμίσουμε ε, ε, το τι ε, και πού πρέπει να δράσουμε και να ενεργήσουμε. Αναμφίβολα πρέπει να επιμείνουμε για τα μέσα ε, ε, αντιμετώπισης και έχουν ήδη αναφερθεί και αναφέρομαι και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Ευρωπόλ που έχουν όλες τις δυνατότητες για να μπορέσουν να εκριζώσουν το πρόβλημα. Και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια όλοι συζητήσαμε σε αυτό το θέμα Και είπαμε ότι έπρεπε όσο γίνεται πιο γρήγορα να κλείσουν οι διαπραγματεύσει για αυτά τα σημαντικά όργανα. Εδώ δεν μπόρεσα να κλείσω αυτό το θέμα γιατί υπήρχαν κάποια... μάλλον να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες λόγω ότι το έπρεπε να είμαι σύντομη αλλά και είναι σημαντικό να ε, καταπολεμηθούν οι απάτες και αυτό προς το υπερφέρων της Ένωσης. Μάλιστα το συζητάμε αυτό και στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, στην οποία επίσης συμμετέχω και για την οποία είμαι, είμαι βέβαια ότι η Κομισιόν πρέπει να υποβάλει οδηγία, πράγμα το οποίο έχουμε ζητήσει επανελειμμένω εδώ στο Κοινοβούλιο, γιατί πιστεύω πως η συμβολή που μπορεί να γίνει από τους ε, ε, πληροφοριοδότες για την ε, αντιμετώπιση των απατών και τη προστασία των συμφερόντων της Ένωσης είναι πολύ σημαντική. Και εγώ ίδια θα υποβάλω τροπολογίες στην ίδια μου την έκθεση ώστε να βελτιωθεί. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Κατερίνα. Ο Τόμας είναι ο σκιώδης του Λαϊκού Κόμματος. Ε, ευχαριστώ πολύ Καταρίνα. Ευχαριστώ πολύ για την ε, εισήγησή σας και ευχαριστώ, συνεργάζομαι μαζί σας για την έκθεση αυτή. Έχω μεγάλο σεβασμό για τα όσα έχετε διπράξει στον αγώνα κατά της καταπολεμήσεως, ε, κατά, συγγνώμη, κατά των απατών. Για μένα προσωπικά η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ενώσεως είναι ζήτημα κέρια σημασίας και παρά την αντίσταση χωρών μελών που δεν αποδίδουν πάντοτε την ε, αρμόζουσα προτεραιότητα στα θέματα αυτά. Η παρούσα Επιτροπή κατάφερε τα τελευταία χρόνια να ε, σημειώσει πολλές επιτυχίες. Η έκθεση λέει, ή θα λέει πιθανότατα, ότι η έκθεση δεν έχει επιτελέσει επαρκή πρόοδο τα τελευταία χρόνια και ιδίως λόγω της απουσίας πλαισίου για την καταπολέμηση απατών, διαφθοράς ε, νομιμοποίησεως ε, παρανόμων εσόδων και ούτω Είναι ανεπαρκή τα εργαλεία, οι μηχανισμοί που έχουμε στη διάθεσή μας και ανίκανα να προσφέρουν επαρκή προστασία στα οικονομικά συμφέροντα της Ενώσεως. Η εισαγωγή της οδηγίας PIF που ακόμα δεν ολοκληρώνεται από το Συμβούλιο, από τις χώρες μέλη. Θα επιτρέψει ωστόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιώσει τον αγώνα κατά των απατών και να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών. Η οδηγία PIF υποτίθεται ότι θα είναι ο πυλώνας πάνω στον οποίο θα μπορέσουμε να βασίσουμε το περίπλοκο οικοδόμημα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ενώσεως, ιδίω για την απάτη σε βάρος του ΦΠΑ. Κάθε εβδομάδα βλέπουμε πλήθος ε, υποθέσεων ε, στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, συλλήψεις απαταιώνων σε χώρες μέλη και ούτω καθεξής. Κάτι που δείχνει ότι ο ΦΠΑ πρέπει να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας PIF. Οι απάτε σε βάρος του ΦΠΑ συχνά σχετίζονται και με άλλες εγκληματικέ δραστηριότητες. Είναι πάντως προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών να καταπολεμήσουν τις απάτες αυτές. Ένα άλλο θέμα που δεν ανέφερε η Καταρίνα, που νομίζω όμως ότι πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι η οδηγία πίφθα προστασία των οικονομικών σφαίρων τη Ένωση, δηλαδή, θα πρέπει να εφαρμοστεί το δυνατόν ταχύτερο. Πολλέ είναι οι χώρες εκείνε μέλη που αντιμετωπίζουν σημαντικότατα ελλείμματα στου προπολογισμού του, δημοσιονομικά ελλείμματα δηλαδή. Και κανένα δεν μπορεί να υπολογίσει πόσα χρήματα χάνουν. Επειδή ακριβώς δεν καταπολεμούμε την απάτη όλοι μαζί. Καθώ και άλλε εγκληματικέ δραστηριότητε. Η οδηγία αυτή, η οδηγία PIF, θα αποτελέσει τον πλέον χρήσιμο μηχανισμό για να καταπολεμήσουμε τι απάτε αυτέ. Ευχαριστώ πολύ. Χουάν Φερνάντο, εσύ. Ευχαριστώ. Ασφαλώς και θέλω και πάλι να επαναλάβω την υπόθεση αυτή των εκκρεμών φακέλων ενώπιον του Συμβουλίου που περιλαμβάνουν και την οδηγία PIF, την οδηγία δηλαδή προστασία οικονομικών συμφερόντων, μέσω του ποινικού δικαίου που έχει κολλήσει στο Συμβουλίο το οποίο δεν κατανοεί τον ρόλο μας ως συνομοθετών. Δεν καταλαβαίνει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, είναι νομοθέτης και στο χώρο του ποινικού δικαίου. Πλήρης νομοθέτης στο ποινικό δίκαιο και ιδίω στην ε, ειδική αυτή περίπτωση για τα θέματα του ΦΠΑ και μετά μάλιστα από την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Βαρίκο δεν υπάρχει καμιά απολύτως αμφιβολία ότι ο ΦΠΑ είναι κέριος φόρος για την ε, εξασφάλιση των εσόδων του προπολογισμού της Ένωσης. Βεβαίω και για τις χώρες μέλη, αλλά ένα μερίδιο του ΦΠΑ καταλήγει στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Είναι λοιπόν κέρια σημασία για τη χρηματοδότηση των πολιτικών της Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να προστατευθεί ο ΦΠΑ απέναντι σε υποθέσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΦΠΑ, αναέτους. Και πάλι όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Συμβούλιο δεν επιδεικνύει καμία προθυμία ή διάθεση να συμβαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά φακέλους που εξυπηρετούν την επίδευση των στόχων που καταστρώνει η συνθήκη λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω για την δικαιοσύνη και ασφάλεια. Και δεν μιλώ μονάχα για την οδηγία ΠΙΦ, ούτε μόνο για τον κώδικα προξενικών θεωρήσεων, αλλά και τόσα άλλα θέματα. Όπου δεν ε, ασκείται καμιά πολιτική, δεν ασκείται καμιά νομοθετική δραστηριότητα, διότι τελικώς το Συμβούλιο είναι ο ελίπων κρίκος στον μηχανισμό της, ε, ε, στους μηχανισμούς μάλλον της Ένωσης. Σας ευχαριστώ Χωάν Φερνάντο και Κατερίνα. Πραγματικά σημαντική γνωμοδότηση. Ευχαριστώ και εσένα Τόμας. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών 25 Οκτωβρίου. Με την άδεια λοιπόν των συναδέλφων τώρα Ας έρθουμε στο 27, το οποίο κανονικά ήταν για αύριο στις 12 και 15. Δηλαδή πρόκειται για, για τον τριμερή διάλογο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. και για την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 475-2002. Θα παρακαλέσω την κυρία Χόλμαϊρ, η συγκίτρια να αναπτύξει το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που είστε και τόσο ευέλικτος ε, στο θέμα της σημερινής διατάξεως. Και πρώτα οι συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διεξάγονται σε ήρεμο κλίμα. Το Συμβούλιο ήδη έχει δεχτεί ορισμένες θέσεις και του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά θέματα όπως για παράδειγμα της εξασφάλισης του ότι στο ζήτημα της προπαγάνδας δεν θίγεται το ζήτημα της έκφρασης προσωπικής άποψης και αυτό να περιληφθεί στο κείμενο. Εξάλλου, σε πλείονα θέματα έχουμε σημειώσει σημαντική προσέγγιση με το Συμβουλίο, όπως για παράδειγμα στο Receiving Training, ή σε ζητήματα recruitment ή σε ζητήματα ιστοσελίδων, όπου ευτυχώς το Συμβούλιο έχει ε, συγκρίσιμη θέση και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί τους. Μένει τώρα ε, για το θέμα των θυμάτων, όπου εκεί έχουμε επιτύχει ήδη ένα πρώτο βήμα προόδου σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός ε, κέντρου συντονισμού και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις στις χώρες μελή, σε περίπτωση δηλαδή όπου σημειώνεται μια επίθεση να έχουν γίνει οι προετοιμασίες ώστε να μπορούν ε, να παρασχεθούν βοήθειες και στα θύματα και όχι να σκέπτεται κανείς μονάχα τους δράστες ε, για την αντιμετώπιση ε, τραυμάτων, ασθενειών κλπ. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα πάντοτε προκάλεσε δυσχέρειες. Δηλαδή όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν ασφαλισμένοι, δηλαδή τα θύματα δηλαδή, δεν ήταν αυτονόητο ότι θα ε, τους παρασχεθούν οι απαραίτητες βοήθειες και η απαραίτητη θεραπεία στη χώρα όπου συνέβη το ε, γεγονός. Άρα πρόκειται και για τον ορισμό του θύματος, επίσης για την ψυχολογική ε, παρακολούθηση των θυμάτων μέσα στα πλαίσια των διαφόρων συστημάτων αλλά και της δικής τους χώρας και της ε, παροχής θεραπείας σε ψυχολογική θεραπεία σε θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων, μπορέσαμε να πείσουμε το Συμβούλιο ώστε αυτό είναι πρόθυμο και σε νομικά θέματα και σε ό,τι αφορά δηλαδή την ποινική διαδικασία αλλά και σε ό,τι αφορά ζητήματα αποζημιώσεων επίσης παροχής πληροφοριών και της ενημέρωσης των συγγενών και τις επαφές μεταξύ νοσοκομείων όπου εδώ ε, σημειώθηκε ένα σημαντικότατο πρόβλημα στο Βέλγιο διότι οι συγγενείς είχαν απελπιστεί, δεν μπορούσαν να βρουν που ε, βρίσκεται ο ανθρωπός τους, σε ποιο νοσοκομείο. Εκεί όπου το Συμβούλιο δεν ε, δέχεται να προχωρήσει είναι να χρηματοδοτήσει συνήγορο για κάθε ένα από τα θύματα. Εκεί το Συμβούλιο έχει στυλώσει τα πόδια και δεν θέλει. Τρεις χώρες μέλη έχουν τον θεσμό αυτό, οι υπόλοιποι δεν θέλουν. Δεν μας βοηθεί λοιπόν πολύ η στάση αυτή. Έχω τον φόβο λοιπόν ότι το Συμβούλιο σε αυτό το θέμα θα παραμείνει πολύ σκληρό. Από την άλλη μεριά πάντως οι συνομιλίες προχωρούν σε άλλα κρίσιμα θέματα. Φαίνεται καθαρά μια διάθεση κινητικότητας από πλευρά του Συμβουλίου. Ελπίζω λοιπόν στις επόμενες συνεδρίες να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες στέρεες συμβαστικές λύσεις όπου να περιληφθούν και οι δικές μας θέσεις αλλά βεβαίως και κάποιες του Συμβουλίου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι πάντοτε φάνηκε πρόθυμη να συμβιβαστεί και μάλιστα ε, συνέρευαν ενεργά και δραστήρια. Ευχαριστώ λοιπόν την Κομισιόν για τον πολύ ε, σημαντικό διαμεσολαβητικό της ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ Μόνικα και η ε, κυρία Τσινίτσι είναι ε, η συγγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κλώδη και ευχαριστώ τη Μόνικα που όντως ανέλησε τη δουλειά που κάναμε μέχρι και χτες ε, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Πρέπει να πω πως όντως το κλίμα που έχει εγκαθιδρυθεί είναι ένα κλίμα ανοιχτό σε συζήτηση και έχουν σίγουρα γίνει κάποιες ε, προσεγγίσεις σε σχέση ε, με τις προτάσεις που κάναμε ε, και στον τριμερή διάλογο. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμβιβαστικές λύσεις όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για αυτές τις πτυχές που δουλεύαμε. Υπάρχει βέβαια αυτό το θέμα το περίπλοκο και δύσκολο της στήριξης δηλαδή στα θύματα. Ε, είναι σίγουρα θετική η ιδέα του κέντρου συντονισμού για τη στήριξη μέσω τέτοιων, ε, τέτοιων ε, κέντρων στήριξη στα θύματα. Το είχαμε πει όμω, είχαμε πει ότι έπρεπε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα γιατί τα θύματα των εγκλημάτων αυτών είναι όλος ο κόσμος, είναι όλοι οι πολίτες, είναι πολίτες που πληρώνουν, διότι τα θύματα ε, είναι οι πολίτες που πληρώνουν τις δράσεις τις τρομοκρατικές που γίνονται κατά του κράτους. Άρα το κράτος έχει το καθήκον να στηρίξει αυτά τα θύματα. Το πιο, πιο περίπλοκος κρίκος είναι όντως ε, τη στήριξη ε, τον, το νομικό Οικονομική ε, άποψη, γιατί αυτό έχει και έξοδα, έχει δαπάνε, επιφέρει δαπάνε. Το είπε και η Μόνικα σήμερα ότι πρέπει ωστόσο να επιμείνουμε για να βρεθεί μια λύση που να δικαιώνει και από αυτή την άποψη τα θύματα της τρομοκρατίας. Κατά τα λοιπά, ε, πιστεύω πως ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμβιβαστικέ λύσεις ε, θετικέ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπή και την, ε, τη συμβολή τη οποία είναι σημαντική για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια ισορροπία που όλοι επιθυμούμε για αυτήν την ε, οδηγία που είναι τόσο σημαντική. Και θέλω να το πω ακόμη μια φορά. Πιστεύω πως είναι σκόπιμο και απαραίτητο να ορίσουμε και να κλείσουμε μάλλον όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ. Thank you. Um, and uh, Mrs. Uh, Κυρία Χιμένες Μπεθερίλ. Hola, sí. <coughs> <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, τη Μόνικα Χολμαϊέρ, για το έργο της, την έκθεση αυτή, που είναι αναγκαία προκειμένου να αντικατασταθεί ε, το πλαίσιο αυτό και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που ξέρουμε ότι λόγω των νέων μορφών τρομοκρατίας ήταν ξεπερασμένη. Υπάρχει ζωσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο, υπάρχουν ε, τα ταξίδια των τρομοκρατών. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Εξάλλου η τρομοκρατία έχει πάντα και ένα, πολιτική σημαντική διάσταση και ιδεολογική βέβαια που δεν θα έπρεπε, αλλά γι' αυτό και εύχομαι κάθε επιτυχία στην ε, η Συγχαίρω επίσης και τη Μόνικα αλλά και την κυρία Κινίτσι που μιλούν για την υποστήριξη των θυμάτων. Όπως ε, είπαν είναι θύματα και της κατάστασης αλλά ολόκληρη η κοινωνία τελικά επομίζεται και μπορεί κάλλιστα να ταυτιστεί με τα θύματα γιατί θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε Όντω χρειάζεται λοιπόν ε, συντονισμό. Το έχουμε πει και εμεί στη ΛΥΜΠΕ. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πρικοδότηση. Και θέλω να εκφράσω κάποια ανησυχία που ακούστηκε, αλλά την λέω και εδώ πάλι. Από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, ότι στα άρθρα δεν θέλουν να μπει ορισμό των θυμάτων. Τι είναι δηλαδή θύμα τρομοκρατίας. Εμένα με εκπλήσει αυτό. Αυτό που λέει το Σεβούλιο είναι ότι υπάρχει οδηγία για τα θύματα. Ναι, αλλά εκείνη, το ξέρω γιατί εγώ την έκανα, λέει για θύματα οποιασδήποτε πράξης βίας. Σου παίρνουν τη τσάντα, σε τραβάνε. Μιλάει και για αυτά. Άλλο είναι αυτό. Εδώ θέλουμε να υπάρξει ορισμός του θύματος τρομοκρατίας συγκεκριμένα όπως ε, το έχουμε κάνει για άλλα θύματα, θύματα σωματεμπορίας για παράδειγμα. Για άλλα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να υπάρξει αυτός ο ορισμός και όπως λέει και η Μόνικα, ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά είναι σημαντικό γιατί όταν έγιναν αυτά που έγιναν στον Πατακλάν, εγώ ήρθα σε επαφή με τη μητέρα ενός νέου που σκοτώθηκε εκεί, που ήταν από τη Γρανάδα, και τι ήταν το πρώτο. Το πρώτο που σου λένε είναι πήγαινε και απευθύσου σε έναν δικηγόρο. Αυτή ήταν Ισπανή, η μητέρα του παιδιού Ισπανίδα. Δεν έχει ιδέα τι ισχύει στην Γαλλία. Φτάνοντας στη Γαλλία είχε αυτό το πρόβλημα. Το πρώτο βήμα είναι να πάει κάποιος σε δικηγόρο για να ενημερωθεί για το τι ισχύει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει και αυτός ο ορισμός και ότι γενικά είναι περίπλοκο το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο. Σε ευχαριστούμε, Τερέσα. Γι' αυτό το θέμα θέλετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Γι' αυτό το θέμα θέλω να μιλήσω, λέει κυρία Μακοβέη, και είμαι σκιώδης εισηγήτρια από το ECR. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τη Μόνικα και όλους τους άλλους που έχουν ε, δουλέψει τόσο σκληρά για αυτή την υπόθεση. Ο τριμερής διάλογος όντως πρέπει να προχωρήσει. Και θέλω να αναφερθώ και εγώ σε αυτά τα κέντρα συντονισμού στις χώρες μέλη. Πιστεύω και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικά γιατί αν ε, λάβει χώρα μια τρομοκρατική επίθεση, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ένα μέρος, ένα κέντρο που συντονίζει όλα όσα συμβαίνουν. Ακόμα και για την μελλοντική βοήθεια που θα θελήσουν να αναζητήσουν κάποια θύματα που δεν έχασαν τη ζωή τους, αλλά είναι θύματα. Συνεπώς όλα αυτά πρέπει να συντονίζονται σε ένα σημείο μόνο στην κάθε χώρα μέλος. Βέβαια, αν συμβεί σε περισσότερε από μία χώρα πρέπει να συνεργάζονται και μεταξύ τους. Το λέω γιατί χτες είχαμε συζήτηση ε, για οδηγία, για νομική αρρωγή. Στις χώρες μας υπάρχει ένα σύστημα νομικής αρρωγής, γι' αυτό δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να μπει στο κείμενο. Στι χώρε μας υπάρχει αυτό το σύστημα νομικής αρρωγής. Όποιο δηλαδή πάει στο δικαστήριο θα το χρησιμοποιήσει. Αλλά κάθε χώρα όπου λαμβάνει χώρα κάποια τρομοκρατική επίθεση θα θέλει να αποζημιώσει τα θύματα και να τα βοηθήσει. Δεν πρέπει να υπάρχουν τεράστιες δίκες, να κρατάνε δεν ξέρω εγώ πόσο χρόνο για να αποφασιστεί ε, τι βοήθεια θα πάρουν. Αυτές τις απόψεις είχα να σας μεταφέρω. Θέλω επίσης να πω ότι πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την υπόθεση όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά και όλους τους φακέλους που έχουμε για θέματα ασφάλειας. Και μην βλέπουμε το Συμβούλιο σαν, πώς να το πω, κάποιον που είναι εναντίον μας. Εδώ δεν είμαστε σε αγώνα μεταξύ μας. Έχουμε τέτοια συμφέροντα να υποστηρίξουμε και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. σε ευχαριστούμε πολύ. 20 Οκτωβρίου θα είναι ο επόμενος τριμερής διάλογος. Η κυρία Χολμάγερ τώρα για να για τις καταληκτικές παρατηρήσεις, αλλά συγγνώμη κύριε Χόλμερ, δεν σε είχα δει Κορνέλια, ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Δεν σε είδα. Ναι, δεν είδα ότι σε στο λόγο. Και είσαι σκιώδης για την ΚΟΕ, ναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, τόσο ήσυχα κάθεσαι εκεί. Συγγνώμη. Παρακαλώ, έχεις το λόγο. Α, φίλε Κλόντ, εδώ βρίσκομαι πράγματι. ορισμένα θέματα. Πρώτον, το πρόβλημα των θυμάτων. Πραγματικά ακαθόδες. Συμφωνώ με τα όσα δήλωσε η σκιώδη συγγήτρια σοσιαλιστών και δημοκρατών. Πρόκειται για ειδική κατηγορία θύματα, έτσι δεν είναι. Ήδη επενδύουμε πάρα πολύ σε μέτρα κατά της τρομοκρατίας. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν και εδώ στην προστασία των θυμάτων. Και η συζήτηση για τον συνήγορο είναι, πώς να πω, λίγο δυσδιάκριτη, διότι βεβαίως πάντοτε κάποια θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων ψάχνουν να βρουν έναν συνήγορο ή συνηγόρους πάντως από ένα δικηγορικό γραφείο. Είναι συχνό αυτό το φαινόμενο. Και έχει καλώς. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ποτέ σε κανέναν ε, να ζητήσει τη βοήθεια συνηγόρου. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που νομίζω ότι οι χώρες μέλη πάνε να βασιστούν σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Και κουράζουν τελικώς με τα επιχειρημάτά τους. Εάν κάποιος επιθυμεί να ζητήσει συνήγορο, να μπορεί να έχει το δικαίωμα να το κάνει. Άλλοι θα κάνουν άλλα πράγματα. Έχει κανός. Το να παρεμβαίνουμε στο δικαίωμα του καθενός να ζητήσει τη βοήθεια συνηγόρου δεν είναι σωστό. Αυτό που είναι σημαντικό για τα θύματα ε, πρέπει να του επιτρέπετε. Το άλλο θέμα είναι, μιλήσατε, συζητήσατε για το αν είναι ποινικό αδίκημα, ε, τρομοκρατική επίθεση, όχι, ε, δεν μπορούμε να το διευκρινίσουμε ίσως ικανοποιητικό, με ικανοποιητικό τρόπο. Εγώ έχω πει αλλού πολλά άλλα πράγματα για το ζήτημα τη προπαγάνδα και τη τρομοκρατίας. Τι είναι προπαγάνδα και τι δεν είναι. Όλα αυτά είναι δύσκολα. Υπάρχουν και πολλές γκρίζε ζώνες. Ε, αν εξετάσουμε τον ορισμό, τα έχω πει αυτά και άλλε φορές, είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι είναι λογική κατά τα άλλα οι ορισμοί και μπορούμε να πούμε όντω ότι ε, οι λύσεις αυτές προτείνονται μπορούν να γίνουν δεκτέ. Και ολοκληρώνω λέγοντα ότι και εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια που πραγματικά διεξάγει συζήτηση μαζί μα και βρίσκω ότι η πορεία που ακολουθεί είναι ορθή και εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Ευχαριστώ Κορνηλία. Μόνικα παρακαλώ εσείς για να ολοκληρώσετε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ με τη σειρά μου τις και όλες τις που είναι βεβαίως παρούσες πάντοτε σε όλες τις ε, συναντήσεις και μάλιστα ε, μας επιτρέπει αυτό να συζητούμε πολύ διεξοδικά και να βελτιώνουμε έτσι διαρκώς τις θέσεις μας. Έχω τρεις παρατηρήσεις τώρα. Πρώτη για το θέμα των θυμάτων. Το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο, και αυτό το βρίσκω θετικό, να δεχθεί τον ευρύτατο δυνατό ορισμό του θύματος. Δηλαδή το θύμα θα ορίζεται, μάλλον από τον ορισμό αυτό θα προκύπτει, θα απορρέει και το ποια δικαιώματα έχει το θύμα και έχουν δεχθεί επομένως εδώ και την οικογένεια να ε, ενταχθεί. Άρα δηλαδή το Συμβούλιο δεν περιορίζει τον ορισμό του θύματος και συμπαρατάσσεται μαζί μας. Αυτό που δεν επιθυμεί να κάνει το Συμβούλιο είναι να βάλει μια ιεράρχηση των θυμάτων. Να πει ότι το θύμα της τρομοκρατίας είναι, αξίζει κάτι περισσότερο από ένα θύμα ενός βιασμού για παράδειγμα. Ε, αυτό είναι βέβαια πολύ δύσκολο θέμα. Με τον δικό μας ορισμό ότι τα θύματα αυτά είναι θύματα διότι η επίθεση στρέφεται κατά του κράτους. Τα συζητήσαμε αυτά και με την Καταρίνα. Συνεχίσουμε να το συζητούμε αυτό. Το δικαίωμα τώρα συνηγόρου έχει ήδη γίνει δεκτό, διότι ο καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει τη σύνδρομη συνηγόρου. Το ερώτημα είναι μόνο ότι η οι χώρες μέλη θέλουν να περιορίσουν αυτή τη δικαστική αρρωγή μόνο στο επίπεδο που την προσφέρουν και εντός της επικρατείας τους και όχι παραπάνω. Ωστόσο οι χώρες μέλη δέχονται ότι η συνήθις δικαστική αρρωγή, δηλαδή το, ε, ε, η, χρηματοδότηση συνηγόρου μέχρι ενός επίπεδου είναι ε, αποδεκτή. Αυτό έχει γίνει δεχτό λοιπόν από τις χώρες μέλη. και αποζημιώσεις το ίδιο. Θα περιληφθούν δηλαδή και οι απαιτήσει ε, για αποζημιώσεις στην οδηγία. Και η ιατρική παρακολούθηση, παροχή δηλαδή ιατρικών ε, φροντίδων και αυτή. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συμφωνηθεί. Πρόκειται τώρα μονάχα για το επίπεδο εισοδήματος από το οποίο και μετά έχει δικαίωμα κανείς να ζητήσει κρατική χρηματοδότηση. Δικαίωμα συνηγόρου το έχουν όλοι, δεν αφισβητείται από καθέναν. Ήθελα να τα πω αυτά ε, διευκρινιστικώς. Τώρα για το θέμα της προπαγάνδας. Έχει εισαχθεί πολύ αυστηρός ορισμός δεν θέλουν να φύγεται με κανένα τρόπο η ελευθερία έκφρασης απόψεως και με παραδείγματα ακόμη, διότι θεωρούν ότι αυτό μπορεί να παράγει τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν θέλουν λοιπόν να υπαχθεί αυτό στην οδηγία. Μονάχα πράξεις οι οποίες εξυπηρετούν την προπαρασκευή τρομοκρατικών υποθέσεων και αυτές βεβαίως πρέπει να αποδεικνύονται. Το κείμενο λοιπόν εκεί στο σημείο αυτό είναι αρκετά καθαρό και στην αιτιολογική έκθεση περιλαμβάνεται επίσης το Συμβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή είχαν και αυτοί παρόμοιες επιφυλάξεις όπως εμείς, ότι οι ορισμοί είναι κάπως υπερβολικά γενικόλογοι, μπόρεσαν λοιπόν να συνεννοηθούν μαζί μας και να συμφωνήσουμε, ώστε να περιληφθεί μάλιστα και ειδική παράγραφος και για τον πάροχο υπηρεσίας, ότι ο πάροχος υπηρεσίας δεν είναι υπεύθυνο για την μεταφορά της ε, σχετικής ειδήσεως. Από την άποψη αυτή, δόξα τω Θεώ, εγώ, έχουμε προχωρήσει αρκετά και το Συμβούλιο έχει προσεγγίσει την θέση μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι για την ε, πραγματικά ε, σημαντικότατη συνδρομή των σκιωδών εισήτριων. Ευχαριστώ, Μόνικα. Ολοκληρώνεται το δεξίτηση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ όλους για την ευκαμψία που δόξα, δείξατε. Θέμα 16 νομίζω με είπε τώρα ο Πρόεδρος. Όχι, ίσως 10. Η κυρία Γκαμπριέλ, το σύστημα υπάρχει μόνο 10. Για την απαλλαγή υποχρεώσεων ε, προξενικών θεωρήσεων ε, ορισμένων χώρων, έξι συνολικά, όπως η η νησιά Μάρσαλ και άλλα. Η κυρία Γκαμπριέλ ε, έχει αναλάβει το θέμα αυτό. Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν να ταξιδεύουν οι πολίτες των χωρών αυτών χωρίς προξενικές θεωρήσεις και βεβαίως προβλέπονται αμοιβαία, ε, αμοιβαία η δυνατότητα Ευρωπαίων πολιτών να ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτε σε επικράτηση των χωρών αυτών για ένα, μια περίοδο μάλλον μέχρι 90 ημερών. Κυρία Γκαμπριέλ, έχετε το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα σας παρουσιάζω τις εκθέσεις αυτές που έχουν να κάνουν με το Κυριμπάτι, Μικρονησία, Κιμπαλού, Νίση Μάρσαλ και Νίση ε, Σολομόντου. Είναι από τις 10 χώρες που πέρασαν από τον Ανατολικό κατάλογο στο θετικό κατάλογο του 539 του 2001 και θέλω να επενθυμίσω τα πλαίσια για την τροποποίηση του κανονισμού. Υπήρξαν διμερώς συζητήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής με όλες αυτές τις χώρες για να καταλήξουν στην απόφαση μη υποχρέωσης ε, θεωρήσεων προσωρινά. Τώρα, εμείς πρέπει να συμφωνήσουμε για το αν αυτό το προσωρινό θα γίνει μόνιμο. Η διαδικασία δεν προβλέπει τροπολογίες, οπότε πρέπει να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την μονιμότητα αυτού του μέτρου. Ποια είναι τα επιχειρήματα τώρα στο σχέδιο έκθεσης. Πρώτον, η προστιθέμενη οικονομική αξία των συμφωνίων αυτών. Είναι το πρώτο στοιχείο που εγώ θέλησα να υπογραμμίσω στην αιτιολογική σκέψη. Ότι οι συμφωνίες δηλαδή αυτέ θα ανοίξουν οικονομικέ δυνατότητε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τι τρίτε χώρε είτε πρόκειται με περισσότερο τουρισμό, είτε με την διευκόλυνση ε, ταξιδιών για τους ε, ενδυνάμει επενδυτές. Στηρίζονται επίσης και δύο παράλληλες οικονομικές διαδικασίες. Πρώτον, η ανάπτυξη του τουρισμού για κάποια από τα νησιά αυτά, Κυριμπάτη και Μικρονησία για παράδειγμα, και διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Εταιρικής Οικονομικής Σχέσης με 13 χώρες του ειρηνικού, μεταξύ των οποίων και αυτές που εξετάζουμε σήμερα. Η κινητικότητα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για τη Συμφωνία εταιρική Σχέσης, προκειμένου να υπάρχουν αμοιβαία ωφέλη. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο κατά τη γνώμη μου είναι η πολιτική και συμβολική αξία των συμφωνιών αυτών. Σήμερα οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα παραπάνω βήμα συγκεκριμένο στην ε, ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ε, χώρες του ειρηνικού που συμμετέχουν στις χώρες ΑΚΕ. Είναι και ένα επιπλέον ε, μέσο για να εντατικοποιηθεί ο πολιτικός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές ελευθερίες, την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος και έτσι μπορούμε να έχουμε και πιο ενισχυμένες οικονομικές σχέσεις. Στα πλαίσια των συμφωνών αυτών θα έχουμε επίσης μια παραπάνω ευκαιρία να συνεχίσουμε και τον πολιτικό μας διάλογο με τις χώρες ΑΚΕ για ζητήματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιπλέον, μην ξεχνάμε σε τι βαθμό η εξαίρεση από την υποχρέωση θεωρήσεων είναι σημαντική για τους πολίτες, για τον τουρισμό, για όσους θέλουν να επισκεφθούν τις οικογένειές τους. Οι συμφωνίες ε, αυτές ενισχύουν την επαφή, την πιο στενή επαφή μεταξύ των λαών και ενισχύει και τη Συμφωνία Κοτονού για τους πολίτες. Τρίτον, στην έκθεσή μου υπογραμμίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ε, για την ασφάλεια των χωρών μας. ...και όλες αυτές τις χώρες δίνουμε την ε, απαλλαγή από τη θεώρηση για βραχίας διάρκειας παραμονή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παραμένουν παράνομα στις χώρες μας. Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Εξάλλου υπάρχει το άρθρο 13 της Συμφωνίας ε, Κοτονού που μιλάει για την επανεισδοχή στην περίπτωση που υπάρξουν τέτοιοι ε, παράνομοι στις χώρες μας μέσα στα διάφορα κριτήρια βέβαια, λέμε ακόμα και όταν αρχίσει να ισχύει η συμφωνία αυτή θα πρέπει να φροντίζουμε να τηρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό του 2014 που είναι ανθρώπινα δικαιώματα και αμοιβαιότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών ανεξαρτήτως καταγωγής. Τέλος, επιμένω και πάλι για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάληξη της συμφωνίας αυτής. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η εφαρμογή τέτοιων συμφωνιών απαλλαγής υποχρέωσης θεώρησης φόσον το Κοινοβούλιο δεν έχει αποφανθεί, δεν είναι σωστό. Γιατί έτσι θέτει υποαμφισβήτηση τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με ξέρετε. Ζητάω λοιπόν από, τη, από να αποφασίσουμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πώς θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως τους συναδέρφους και κυρίως τους κοιόδες εισηγητές για τη βοήθειά τους και προτείνω σύντομα να εγκρίνουμε τις πέντε αυτές εκθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκαμπρίλ. Ποιος θέλει τον λόγο. Α, Σκιώδης, εισηγήτρια από το Άλντε, έτσι. Παρακαλώ. Κυρία Ισμανόβα, Ισμανόβα. Εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Γκαμπριέλ, για την εργασία της σε αυτό το φάκελο, καθώς εξ ονόματος της ομάδας Άλντε θα ήθελα να τονίσω ότι η άνευ θεωρήσεων Ε, μετακίνηση ωφελεί τους πολίτες των τρίτων χωρών αλλά και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τηρούνται τα κριτήρια. Αυτό ενισχύει το διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση. Ε, θέλω να τονίσω και πάλι την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπίζεται ως ισότιμος νομοθετη, νομοθε, ε, όπως λένε άλλωστε και οι συνθήκες. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιμάνοβα. 18 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και Ευχαριστώ κυρία Γκαμπριέλ. Σημείο 17 νομίζω, γιατί έχουμε τόσο πολύ ανακατέψει τη μυρίσια διάταξη που πια δεν ξέρω. Εφόσον δεν με διορθώνετε, πάω στο 17. Εδώ έχουμε ακόμα μια παρουσίαση Όσον αφορά την αναθεώρηση ακόμα μιας νομοθεσίας. Ε, δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Έχουμε τον κατάλογο ε, υπηκών τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. 7 Ιουλίου είχαμε μια ψηφοφορία εδώ. Δώσαμε εντολή στον εισηγητή και στη διαπραγματευτική ομάδα να ξεκινήσει διαπραγματεύση με το Συμβούλιο για την Επιτροπή ε, εν ώψη συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Θα θυμάστε τι προσπάθειε που καταβλήθηκαν να προχωρήσουμε με αυτό το θέμα γρήγορα και στην πρώτη έκθεση στην Λίμπε έγινε στι 31 Οκτώου. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντία Δεμέρα Ε, για να μας πει που βρισκόμαστε. Έχετε το λόγο. Sí, muchas gracias, señor presidente. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, όντως, ε, συμμερίζομαι και επαφάνω τα όσα είπατε. Θέλω να σας πω ότι θα ήθελα να σας ενημερώσω για το ποια κατάσταση βρισκόμαστε στην έκθεσή μου σε σχέση με τον ε, ε, μηχανισμό αναστολής. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους του Σκιώδης γιατί με ε, στήριξαν ομόφωνα σε αυτή τη τόσο περίπλοκη τεχνική ε, έκθεση που και από πολιτικές άποψεις είναι ευαίσθητη και φυσικά να ευχαριστήσω την γραμματεία να τονίσω και να δείξω την επαγγελμα... τον επαγγελματισμό των ε, της γραμματείας. Να δώσω κάποιες ημερομηνίε για να καταλάβετε ε, πού βρισκόμαστε στην πορεία εξέταση αυτή τη νομοθεσία. 26 Μαΐου ανέλαβα την έκθεση. Υπέβαλα την πρώτη στις 15 Ιουνίου. Ψηφίσαμε στην ΛΥΜΠΕ για την διαπραγματευτική εντολή στις 4 Σεπτεμβρίου. Ο πρώτος τριμερής έγινε στις 6 Ιουλίου. Η πρώτη ε, επαφή με τον πρέσβη εκπρόσωπο της Σλοβακίας στις 27 ε, Σεπτεμβρίου. Με... Έπρεπε να κάνουμε, να πω ότι από τον πρώτο τριμερή μέχρι την πρώτη επαφή με τον πρέσβη πέρασαν 83 μέρες. Αυτό με ενοχλεί να που σα το λέω, αλλά έτσι έγινε. Ε, και αυτέ οι ημερομηνίε δείχνουν ότι το Κοινοβούλιο εντατικά εργάζεται ώστε να ξεβρεθεί η συμφωνία. Κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω εξίσου για το Συμβούλιο. Ε, μας πίεσαν, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, γιατί εκφράζει πολύ καλά την ε, πραγματικότητα και ξεκολουθούν να μας πιέζουν με κάθε μέσο ε, Όμως αυτό δεν αντιστοιχεί με την ε, καθημερινή ε, άνεση προτάσεων που είναι σε θέση να οδηγήσουν στην εξέβρεση μιας διοργανικής συμφωνίας και πρέπει μάλιστα να τονίσω γιατί ακριβώς αυτό συμβαίνει ότι οι πιέσεις είχαν πολύ συγκεκριμένη χρονική έκτακτη φάση και ειδικά εντάθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Για αυτού του λίγου που λένε ότι το Συμβούλιο είναι το μόνο που κινείται και το Κοινοβούλιο μπλοκάρει αυτή την έκθεση, να σας πω ότι είναι λάθος, Εντελώ λάθος. Αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο έχει υποβάλει τρει συμβιβαστικέ λύσει διαφορετικές για να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Η πρώτη πρόταση, σας θυμίζω, ε, συνίστατο στο ότι προσφέραμε τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός μέσω κοινοποίησης με απλή πλειοψηφία των κρατών μελών, χρησιμοποιώντας αυτό το οποίο συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί τη κατεξουσιοδότηση πράξης. Δε, δεύτερη πρόταση ήταν ότι θέσαμε στο επιτάπητο στη δυνατότητα ανάπτυξης του μηχανισμού χρησιμοποιώντας κατεξουσιοδότηση πράξης μέσω της διαδικ... πήγουσας διαδικασίας. Και η τρίτη πρόταση είναι η ε, ε, κίνηση του διαδικασίας μέσω τριών φάσεων, όπως γνωρίζει πολύ καλά και ο Πρόεδρος, αυξάνοντας την πίεση στο τρίτο μέλος ε, το ενδιαφερόμενο και εξετάζοντας μια μεικτή δράση μέσω εκτελεστικών και πράξεων και πράξεων κατά εξουδότηση, χρησιμοποιώντας το μηχανισμό αμοιβαιότητας. Όμως, το Συμβούλιο δεν άλλαξε ούτε καν ένα γράμμα στην πρότασή του και υπερασπίστηκε αντιμετωπίζεται με τροπολογίε μια πρόταση η οποία είναι παράνομη. Ανακατεύει, αναμειγνύει χωρίς καμία νομική αιτιολόγηση ε, κατεξοδότηση πράξη και πράξει εκτελεστικές. και αυτό δεν, είναι, δεν το λέω εγώ αλλά το έχουν επιβεβαιώσει και οι νομικές μας υπηρεσίες, καθώς και το δικαστήριο. στην απόφαση του 088 κάθετος 14. Και θα το επαναλάβω ξανά και ξανά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια κοινή νομική βάση μέσω των δικών μας νομικών διαδικασιών, διαφορετικών μάλλον νομικών διαδικασιών. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ε, για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα πρέπει να δώσουμε τις ίδιες λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι δικές μας προτάσεις να δώσουν απάντηση στα αιτήματα του Συμβουλίου. Θα ήταν αυτός ένας καλός δρόμος να ακολουθήσουμε ώστε να εξευρεθεί συνένεση και κυρίως οι προτάσεις μας είναι νόμιμες. Θέλω και να προσθέσω δε ότι ότι πρόκειται για εξαιρετική, ε, ότι θα ήθελα να ακούσουμε μάλλον πληροφόρα νέα από το Συμβούλιο και καλό θα ήταν εδώ και την παρουσία της Επιτροπής ε, να ακούσουμε κάτι το θετικό. Από ό,τι φαίνεται η τελευταία μας πρόταση έγινε καλά δεχτή από πλευράς ε, των κατών μελών και θα μπορούσε και να χρησιμεύσει ε, ως βάση για μια μελλοντική συμφωνία. Ε, το Συμβούλιο δε ε, υποσχέθηκε να υποβάλει μια νέα πρόταση πριν ε, την Παρασκευή. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ε, αν όντως συμβεί αυτό, θα, θέλα, θα μπορούσαμε ε, να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες και αν είναι δυνατόν να φτάσουμε και σε συμφωνία γρήγορα. Να κάνουμε δηλαδή και τριμερή διάλογο την ίδια την Τετάρτη. Ε, Πέρα από το θέμα των καταξιοδότησης πράξεων των εκτελεστικών πράξεων, ε, φτάσαμε σε σημαντικέ συμφωνίες ε, στα εξή σημεία. Σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σύστημα παρακολούθησης από πλευρά της Κομισιόν, καθώς και μια πληροφορία που θα ήθελα να σα δώσω και να επαναλάβω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου για την κατανόησή σας και για να τη στήριξή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα περνάμε στο Συμβούλιο και μετά στα κράτη. Ε, στη, συγγνώμη, στους ε, βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, Μπίργκιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται, πρέπει πάλι να υπογραμμίσουμε ότι είναι φυσιολογική νομοθετική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνεται με το δύο συνομοθέτες και σε αγαστή συνεργασία, δηλαδή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και επειδή αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο είναι συνομοθέτες για όλα τα θέματα θεωρήσεων, φυσικά και είμαστε συνομοθέτες για κάθε είδος μηχανισμό αναστολής. Ε, το να αποφύγουμε αυτό και να λέμε ότι δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα είναι γελίο. Εγώ ε, έχω μεγάλο σεβασμό για το συναδελφό Δίας Δεμέρα, τον εισηγητή μας. Και θα πρέπει να πούμε ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, καθώς και ο εισηγητής μας, έκανε ό,τι γινόταν ε, ώστε να κινηθούν ε, ε, τα πράγματα και να προτείνουμε συμβιβαστικέ. Από πλευρά του Συμβουλίου όμως δεν έχει υπάρξει καμία κίνηση. Ε, δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν, μπορούμε να, δεν μπορεί να το δεχτεί την πρότασή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, έχουμε μια πολύ καλή συμβιβαστική για να εξασφαλίσουμε ότι οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο, ε, το Συμβούλιο θα ξεκινά διάλογο με τις χώρες όποτε προκύπτει δηλαδή πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε το, του το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να συμμετέχει όταν αυτό είναι απαραίτητο για να αναστέλλεται η θεώρηση. Ε, ή όποτε, βάση περιπτώσει, προκύπτει θέμα. Γι' αυτό και ελπίζω πραγματικά πως το Συμβούλιο θα κινηθεί επιτέλους ώστε να κλείσει αυτός ο φάκελος ε, με αίσιο πέρας από αυτή της βάσης της συμβιβαστική που έχει υποβληθεί ε, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και με τις, την κατάργηση των θεωρήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προεδρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για τις διαπραγματεύσεις που είχαμε μέχρι τώρα. Έχουμε προχωρήσει όσον αφορά τις διαδικασίες και κάποιες νομικές πτυχές. Πάνω απ' όλα θέλω να συμφωνήσω με αυτό που είπε στα συμπεράσματά του ο κύριος Όταν δηλαδή μιλάει για ενθαρρυντικές εξελίξεις. Όντως. Πιστεύω ότι την τελευταία εβδομάδα περάσαμε σε ένα πιο θετικό στάδιο των διαπραγματεύσεών μας. Και Πιστεύω ότι η πρόταση που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα θα ληφθεί, θα κληφθεί ως βάση για να διακανονιστεί αυτή η υπόθεση. Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω την Επιτροπή σας, τους αξιότιμους ευρωβουλευτές, ότι αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Προεδρίας αυτός ο φάκελος και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να καταλήξουμε σε συμφωνία πράγματι πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον κύριο Τίεφτε Μέρα και την Προεδρία που έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε, παρόλο που δεν είναι πάντα εύκολη συζήτηση με τις καταξιδότηση πράξεις και τις εφαρμοστικές. Συζητήσαμε πράγματι το συμβιβασμό που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή και όπως είπε και η Προεδρία και για μας θα αποτελέσει βάση για τη συνέχεια. Ήδη στην πρόταση αναφέρονταν ότι αν υπάρχουν στοιχεία για την κατάσταση σε μια χώρα για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση θεωρήσεων, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρθει σε διάλογο με τη χώρα αυτή για να δει σε τι βαθμό μπορούν να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Δεν χρειαζόμαστε εφαρμοστική πράξη ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπούμε σε ένα τέτοιο διάλογο. Αυτό το είπαμε και στον τριμερή διάλογο και νομίζω ότι το κατάλαβε το Κοινοβούλιο. Ελπίζω επίσης ότι οι νομικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα μπορέσουν να μιλήσουν μεταξύ τους γιατί είναι δύσκολο να έχουμε κάτι που ο ένας το θεωρεί παράνομο και ο άλλος όχι. Καλό θα ήταν λοιπόν να γίνουν και τέτοιες συζητήσεις, εκ παραλίλου ότι άλλες συζητήσεις γίνουν εν ώψη του επόμενου τριμερής διαλόγου. Οι νομικές υπηρεσίες να συζητήσουν μεταξύ τους αυτά τα θέματα έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε με τον ίδιο τρόπο όλοι. Και να δούμε μήπως τελικά υπάρχει διαφωνία επί της νομιμότητας που δεν θα έπρεπε σε ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Όχι, οπότε περιμένουμε την πρόταση του Συμβουλίου, κύριε Διευθυντεμέρα, την Παρασκευή, σωστά? Θέλετε να σχολιάσετε τίποτα για να κλείσουμε αυτό το θέμα? Το μόνο που θέλω να πω, Πρόεδρε, είναι το εξή. Ε, για λόγους, ε, αν μη τι άλλο, ευγένειες, να ευχαριστήσω για τα τόσο θετικά σχόλια και ευχαριστώ και την κυρία Σίπελ, τον Βλαμίντιρ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ και θα δούμε τι θα γίνει τώρα με το έγγραφο της Παρασκευής. Ωραία. Θα περάσουμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο, περιμένοντας τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι, για την υπομονή σας. Καλύψαμε πολλά θέματα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημείο 18. Απλώς θέλω να σας πω, συνάδελφοι, ότι στις 3 έχουμε την ακρόαση της Επιτροπής μας για τη συνεργασία Σέγγεν, παρόν και μέλλον. Εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Γι' αυτό παρακαλώ να είσαστε εδώ στις 3 ακριβώς για να ξεκινήσει η ακρόασή μας. Έληξε η συνεδρίαση λίγο νωρίτερα σήμερα. Θα τα ξαναπούμε στις 3 για την ακρόαση με θέμα το Σέγγεν.